Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Merci de votre présence. Premier point, l'adoption de l'ordre du L'ordre du jour, s'il n'y a pas de nous le considérons comme adopté. Έχετε την διάταξη, πιστεύω την να μου πείτε αν έχετε κάποια παρατήρηση. στο δεύτερο σημείο της Μάλλον όχι, στο πρώτο, στην έγκριση. Υπενθυμίζω ότι στι 17.30 και 30 ολοκληρώνονται οι εργασίε τη Επιτροπή των Προπολογισμών. 17 και 30 έω 18 και 30, 5.30 με 6.30 το βράδυ, θα γίνει συνεδρία των συντονιστών. Για να συζητήσουμε μια δεύτερη ανάγνωση του προπολογισμού 2010 και του ψήφου που θα τον συνοδεύσει. Και αύριο το πρωί ξεκινούμε από τι 9. και παρακαλώ τακτικά και αναπληρωματικά, αλλά και αναπληρωματικά των αναπληρωματικών μέλη, παράνομα λαθρέα και παρισφρήσαντα, να είναι όλοι παρόντες για τη δεύτερη ανάγνωση. Ανακοινώσεις. Συγχαίρω τον συνάδελφο κύριο Κοτμάνης, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του πριν από μερικές μέρες. Πολύχρονος Κάθε μέρα είστε και πιο νέος. Ένα Και επίσης θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η σημερινή ημέρα έχει ιστορικό χαρακτήρα. Γιατί σημειώνει τη θέση ισχύ της συνθήκης Λισαβόνος. Παραδόξως πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο δεν προτίμησε να χαιρετήσει τη θέση ισχύ επισήμως σήμερα εδώ Στη Λισαβόνα λαμβάνει η χώρα μία τελετή στην οποία μας εκπροσωπεί ο πρόεδρος Μπούσεκ, αλλά το κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες δεν εορτάζει τη θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Πράγμα το οποίο ενδεχομένω ορισμένοι να θεωρούν λυπηρό άνθρωποι ιδιαίτερο όπω ο πρόεδρο Δεάνε, ο οποίο έχει συμβάλει τόσο πολύ στην επεξεργασία του κειμένου, όπω και άλλοι πολλοί που ήταν παρόντες στη συντακτική συνέλευση για το Σύνταγμα, για του ίδιου συντάγματο. για όλου εμά εδώ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερο μέλη τη Επιτροπή των Προπολογισμών, για όλου εμά του πολίτε τη Ευρώπης, είναι η ημέρα αυτή μεγάλη και ας μην την τιμούμε. Μια μεγάλη ιστορική ημερομηνία που θα γραφτούμε ξαγράμματα στην ιστορία της Ευρώπης, αναλόγως βέβαια του τι τύχη θα επιφυλάξουμε εμείς στην συνθήκη αυτή και κυρίως πώς θα χειριστούμε τα δημοσιονομικά θέματα. ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σημειώνουμε τις νέες αρμοδιότητες που μας ε, αναγνωρίζει πλέον ε, η συνθήκη και σε αγαστή συνεργασία εφόσον είναι δυνατόν, με τα άλλα θεσμικά όργανα και σε αντιπαράθεση με τα άλλα θεσμικά όργανα όπου είναι απαραίτητο Όπου δεν υπάρχει λύση θα επιτελέσουμε το καθήκον μας ως οφείλουμε. Και ευχαριστώ εδώ την ε, ε, εκπροσώπηση της Επιτροπής και της Σουηδικής Προεδρίας, μάλλον της Σουηδικής Προεδρίας, την ευχαριστώ ιδιαίτερα που είναι εδώ παρούσα, και όταν έρθει θα καλωσορίσω και τον υποψήφιο Επίτροπο για θέματα προϋπολογισμού, που είναι γνωστός οικείος στα μέλη της Επιτροπής μας, δεν θα τον συγχαρούμε επισήμω βέβαια σήμερα, διότι ο τυπικός, η τυπική πράξη του διορισμού εξαρτάται από εμά και από τις απαντήσεις που θα δώσει στις πολύ σκληρές και δύσκολες ερωτήσεις που θα του υποβάλουμε στη διαδικασία που προβλέπεται για τη δεύτερη ε, εβδομάδα του Ιανουαρίου. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο ενέκρινε η διάσκεψη των Προέδρων για τις ακροάσεις στη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, λόγω των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τους ορισμούς που ανήκουν στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, ε, σημαίνουν εν τέλει ότι κατά μία εβδομάδα ιδιαίτερης, ε, ιδιαίτερου χαρακτήρα, Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου δηλαδή θα προβλεφθεί η διεξαγωγή όλων των ακροάσεων, όλων των υποψηφίων επιτρόπων, ενώπιον όλων των ε, αρμοδίων επιτροπών του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι εφόσον βέβαια όλα πάνε καλά και εφόσον ε, προκύψουν θετικές νομοδοτήσεις από το Κοινοβούλιο για τις υποψηφιότητες αυτέ, αυτές, σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο του Ιανουαρίου. Εάν υπάρχουν προβλήματα θα πρέπει να κληθεί ο πρόεδρος Παρούσο να αλλάξει, να αλλάξει τη σύνθεση της ομάδας του, περίπτωση κατά την οποία θα προβλεφθεί μισή ημέρα για την, ε, στην τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου για να συζητηθούν ε, αυτές οι αλλαγές. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Κατά τα άλλα, υπενθυμίζω ότι η συνεδρίαση αυτή, όπως και οι προηγούμενες, ε, μεταδίδονται μέσω του διαδικτύου. Υπενθυμίζω ότι η σημερινή και η ευριανή συνεδρίαση είναι κατ' ουσίαν αφιερωμένες την διευκρίνηση στρατηγικής μας για τη δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου προπολογισμού 2010 που θα συζητήσουμε ευθύ αμέσω. Για να προσδιορίσουμε στη συνέχεια ότι χρειάζεται διευκρίνηση σε επίπεδο συντονιστών ε, προς το τέλος της ε, συνεδρίασής μας, δηλαδή το απόγευμα, ώστε αύριο να προβούμε στην ψηφοφορία. Σας διανέμουμε ήδη τώρα τα έγγραφα που θα χρειαστείτε για την ψηφοφορία. Και σας παρακαλώ να τα φέρετε μαζί σας και αύριο. Θα τα χρειαστούμε. Για την ψηφοφορία. Θα προσπαθήσουμε να ενοποιήσουμε στο βαθμό του δυνατού τις ψηφοφορίες. Θα σας εξηγήσω αύριο το πρωί πώς ε, ποια είναι η λογική των εγγράφων. Δεν χρειάζεται τώρα να χάσουμε χρόνο με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι το περίπλοκο φυσικά, αλλά καλό θα είναι και ο καθένας να έχει αντιληφθεί τις ε, διαφορές μεταξύ των εγγράφων. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες για τη δεύτερη ανάγνωση που έχουν χαρακτήρα περισσότερο επεξηγηματικό και όχι πολιτικό, αλλά το βασικό είναι να έχετε τα έγγραφα μαζί σα. Και εν τέλει, Θα ήθελα να εξηγήσω να ε, ε, δώσω τα αποτελέσματα από τις συνεδρίες των συντονιστών ε, της προηγούμενης εβδομάδας, όπου κατανεμήθηκαν δύο εκθέσεις, πιθανές νομοδοτήσεις, όσον αφορά την χρηματοδοτική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη χρηματοδότηση των μονάδων υπαριθμών 1 και 4 ε, σχετικά με την πάυση λειτουργίας του σταθμού του Κοσλοντούι. Νομική βάση. Έχουμε συμφωνήσει και έτσι πρέπει να ψηφίσουμε τη χρηματοδότηση του σχετικού κονδυλίου για το 2010. Όμως πρέπει να εγκρίνουμε τη νομική βάση πρώτα, βάση της οποίας δίνουμε γνωμοδότηση, ενόψη της οποίας μάλλον δίνουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή Βιομηχανίας, η οποία θα προσδορίσει μετά και θα προσδοριστεί από αυτήν ο εισηγητής. Για δε την χορήγηση μακροοικονομικής ενίσχυσης στην Ουκρανία συμφωνήσαν ε, οι συνάδελφοι ότι δεν έχει λόγο να γνωμοδοτήσει η Επιτροπή των Προϋπολογισμών και ως εκ τούτου δεν προσδορίζεται εισηγητής. Σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Προετοιμασία της δεύτερης ανάγνωσης του Κοινοβουλίου. Το λόγο έχει ο εισηγητής, συνάδελφος Λάσλο Σούτζιαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είμαι σίγουρος ότι στις διάφορες ομάδες εργασίας ε, οι συνάδελφοι έχουν ήδη κατανοήσει τι συμβαίνει, τι συνέβη μάλλον ε, στην συνδιαλλαγή. Ενδεχομένως όμως καλό θα ήταν να κάνω μια σύνοψη του τέλους της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Όπως γνωρίζετε, ο φετινός προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα, δηλαδή το δεύτερο τμήμα της, του Συμφώνου Ανάκαμψης. 2,9 δις. Δεν είναι καθόλου εύκολο να διαχειριστεί κανείς ένα τέτοιο ποσό χωρίς να επηρεάσει καθόλου τις ήδη υπάρχουσες διαδικασίες και τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Βεβαίως, ε, επ' αυτού το Κοσλοντούι ήταν ένα μικρό πράγμα, αλλά και κάτι ε, καινούριο, το οποίο προστέθηκε στο όλο οικοδόμημα το οποίο οφείλουμε να διαχειριστούμε. Εν τω μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον το, έτσι ώστε να προσφέρει κάτι στον γαλακτοκομικό τομέα λόγω των προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίσαμε σε αυτόν τον τομέα ιδιαίτερο το φθινόπωρο. Και η φιλοδοξία των περισσότερων μεταξύ ημών ήταν να μην ε, έχουμε αυτό το, σχέδιο ανάκαμψης και για τον επόμενο χρόνο. Αλλά βεβαίως δεν ήταν και σαφές εάν θα ήταν δυνατόν να διαχειριστούμε την κατάσταση ε, μέσα στα πλαίσια του 2010 ή όχι. Τέλος, συμφωνήσαμε ότι θα ολοκληρωθεί το ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης το 2010 και δεν θα μείνει τίποτα για την επόμενη χρονιά. Επίσης, και για πρώτη φορά στα πλαίσια του πνεύματος της, Λισαβόνης, της Λισαβόνας το ε, Συμβούλιο δέχτηκε μία επιπλέον βοήθεια 300.000 ε, για τον γαλακτοκομικό τομέα για τους κτηνοτρόφους ε, και αυτό βεβαίως ήταν μια συμβολική αλλά και όχι μόνο ε, κίνηση αναγνώρισης ε, της αξίας του Κοινοβουλίου. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είμαστε νικητές. καταλαβαίνουμε ότι αριθμητικά μπορεί να πρόκειται για ένα μικρό στοιχείο σε σχέση με άλλα, αλλά παρόλα αυτά πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Ε, γιατί και το Συμβούλιο και η Κομισιόν ε, είχε, είχαν αποδεχθεί ε, το θέμα αυτό και δέχτηκαν να βοηθήσουν. Επίσης, η Επιτροπή Απασχόλησης καλοδέχτηκε αυτά τα επιπλέον χρήματα, από τα οποία δεν πήραξαν όμως οποιαδήποτε, οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για μια καλή κίνηση. Τώρα, το απαραίτητο ποσό για την πρώτη χρονιά ήταν 25.000 και έγινε δεκτό το ποσό αυτό. Επίσης, συγγνώμη, 25 εκατομμύρια. Και βεβαίως το Συμβούλιο δέχτηκε το μήνυμά μας όσον αφορά το Big όπου ε, η προσέγγιση ήταν αρκετά εξεζητημένη και πρόκειτο για ε, μία ε, για έναν συνδυασμό ε, γραμμών και λειτουργίας γραμμών του προϋπολογισμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε λίγο μεταξύ του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Και αυτή η θέση όμως έγινε δεκτή από το Συμβούλιο και επομένως είμαστε σε θέση να την διατηρήσουμε στην δεύτερη ανάγνωση. Επίσης, φιλοδοξία μας ήταν να προετοιμάσουμε το διάλογο και τις προπαρασκευαστικές δράσεις έτσι όπως ψηφίστηκαν στην πρώτη ανάγνωση. Και είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε τώρα, κατά αυτή την έννοια, στη δεύτερη ανάγνωση μετά από την συμφωνία ε, με το Συμβούλιο. Όσον αφορά τις πληρωμές, μπορεί κανείς να δει το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Σε αριθμούς πρόχειρους υπολογισμούς. Το Συμβούλιο πρότεινε 120 δις, η πρώτη μας ανάγνωση ήταν 127. Όλοι μας γνωρίζαμε ότι επρόκειτο για μία αύξηση η οποία ήθελε να καταδείξει την πολιτική μας βούληση και θέλαμε να δείξουμε επίσης ότι θέλουμε καλύτερη χρήση, αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη ε, των χρημάτων, των ταμείων ε, των διορθωτικών αλλά και της συνοχής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των κρατών μελών και επομένως ε, θα υπάρξει τροποποιητικός προϋπολογισμός έτσι ώστε να καλυφθούν αυτές οι πραγματικές ανάγκες. Θα δούμε πώς θα το κάνουμε κάθε χρόνο γνωρίζετε βεβαίως καλύτερα από μένα ότι μέχρι τώρα η δυνατότητα αυτή δεν χρησιμοποιήθηκε. Όμως, εάν το 2010 αποτελέσει τη χρονιά όπου θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα και λόγω του ότι μάλιστα παρουσιάζεται μεγάλη καθυστέρηση ε, σε πολλές ε, χώρες, αλλά ε, ε, υπάρχουν και προγράμματα τα οποία έχουν συσσωρευτεί το 2007, 2008, 2009. Είναι αρκετά όρημα και επομένως ε, η ανάγκη πληρωμών στα πλαίσια αυτής της πολιτικής συνοχής είναι ή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει εάν στους, στους, στους συντονιστές συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι μια λεπτή κόκκινη γραμμή και είπαμε ότι τώρα δεν θα ε, κατεβούμε λιγότερο, χαμηλότερα από το προσχέδιο του προϋπολογισμού όσον αφορά την ε, ε, πολιτική συνοχής. Άρα πρέπει να προετοιμάσουμε όλες αυτές τις, τις προπαρασκευαστικές δράσεις εντός των πλαισίων και των γραμμών του προϋπολογισμού. Τώρα να πούμε κάτι για τα μεγάλα νούμερα, τα ψηλά νούμερα στα ποσοστά του GNI. Ένα για πληρωμές, 1,02 σε δεσμεύσεις, σε υποχρεώσεις. Αυτό σημαίνει αν θυμάστε, ε, υπάρχει πάντα μια διαμάχη ανάμεσα στις ε, χώρες μέλη που πληρώνουν και τις άλλες, ε, γιατί αυτές δεν θέλουν ε, ε, προϋπολογισμό πάνω από το 1%. Ε, η Σουηδική Προεδρία όμως έδειξε κάποια ευελιξία, παρουσίασε επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σωστή επιχειρηματολογία και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτό το 1,04 και το 1,02. Όσον αφορά τώρα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης, το ερώτημα ήτο, ποιος θα πληρώσει περισσότερο. Ο πρόεδρος μας, ο κύριος Λαμασούρ, είχε ένα όραμα και βεβαίως ένα καλό επιχείρημα. Δηλαδή ότι για να περικόψει κανείς κάτι, ε, η περικοπή αυτή θα είναι σίγουρα οδυνηρή. Πιο οδυνηρή από το να δώσουν ε, φρέσκο χρήμα, λέει ο μιλητής, στα κράτη-μέλη. Και επομένως, στόχος μας ήταν ότι για μία μείωση του 1 ευρώ, ευρώ από το 1α θα σήμαινε μείωση 2 ευρώ αντίστοιχη. θα έπρεπε ας πούμε να περικόψουμε 81 εκατομμύρια στο κεφάλαιο Α1 συμπεριλαμβανομένου του Κοσλοντούι που από μόνο του είναι 75, 75 και το Συμβούλιο από τον Μηχανισμό Ευελιξίας έδωσε 195 από το περιθώριο του κεφαλαίου 2. Πράγμα που είναι, αν θυμάμαι καλά, 36 εκατομμύρια πάνω από τα προβλεπόμενα. Και επομένως, ο εισηγητής έπρεπε να αποφασίσει και να προτείνει κάτι σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να περικοπούν αυτά τα 81 εκατομμύρια στο 1α. Ακούγοντας και τη γνώμη των συντονιστών, περίμενα ότι, θα, ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα μπορούσε να αποτελέσει ε, την, το κατόφλι αυτής της ε, περικοπής. Δηλαδή να μην ξεπεράσουμε αυτό το όριο προς τα κάτω. Τώρα, εάν αυτές οι περικοπές μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα έστω και μικρό περιθώριο, Κοινή δέσμευση ήταν και κοινή επιθυμία να δώσουμε το 25% στο εργαλείο διευκόλυνσης της μικροπίστωσης. Και τα υπόλοιπα χρήματα να μοιραστούν σε 7 γραμμές οι οποίες είχαν την προτεραιότητα. Όπως ας πούμε η εκπαίδευση, η έρευνα κτλ. Κατανείμαμε τα χρήματα σύμφωνα με ε, ποσοστά της 100 ε, συνδυασμού ας πούμε των γραμμών αυτών με άλλες γραμμές. Και στο τέλος βρήκαμε ότι είχαμε ένα 0,7 ανοιχτό ακόμα και διαθέσιμο. Είχαμε και την στήριξη της Άλντε βέβαια ε, στην απόφαση ότι τα χρήματα αυτά μπορεί να είναι λίγα αλλά παρόλα αυτά ε, θα μπορούσε να δοθεί ένα θετικό μήνυμα, όχι εξαιρετικά σημαντικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα ε, μήνυμα ε, θετικό προς το χρηματοδοτικό εργαλείο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν ότι οι φιλελεύθεροι συμφωνούσαν με την ιδέα και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και ο εισηγητής ήθελε να έχει ευρύτερες συνεργασίες, προτείνουμε ε, να έχουμε αύριο τον ε, χρόνο να αποδείξουμε στο Συμβούλιο και την Κομισιόν ότι μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και ότι θα είμαστε πολύ δυνατοί υπό την συνθήκη της Λισαβόνας. Το ερώτημα είναι ανοιχτό. Δηλαδή, τι θα κάνουμε με το υπόλοιπο από αυτό το περιθώριο λαμβάνοντα υπόψη ότι είναι πάρα πολύ λίγα χρήματα. Βέβαια, η μία άποψη είναι, η μία επιλογή είναι να τα αφήσουμε. Και θα ήθελα να ξέρω την άποψή σα από αυτού. Σω το καλύτερο θα ήταν να τα αφήσουμε. Σα εξηγώ δε ότι ίσω είναι καλύτερα και θα σα πω γιατί. Ακόμα και η γραμματεία Ε, μπορεί να μας δώσει πολύ καλά αποτελέσματα και αριθμητικά στοιχεία, αλλά ξέρετε ότι ε, αλλάζοντας ας πούμε βάσεις δεδομένων, databases, μπορεί ε, να βρει κανείς το διάβολο στις λεπτομέρειες και εμπροκειμένου το διάβολο στα στοιχεία τα οποία βρίσκονται στη μία ή στην άλλη βάση. Επομένως, μιλάμε για μία πάρα πολύ μικρή διαφορά και επομένως μπορούμε ε, να μην έχουμε αυτή την τεχνική προσαρμογή του εισηγητού στην ε, ε, Ολομέλεια και νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν και για τον κύριο Μάνκα και για μένα να αποφύγουμε αυτήν, αυτή την προσαρμογή στην Ολομέλεια. Αυτό βέβαια θα μου το πείτε εσείς τι θέλετε να κάνω. Αλλά ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει μία λύση. Εάν ε, βεβαίως η η Επιτροπή, η μας εδώ, μέσα στη σοφία της, αποφασίσει να βάλουμε ένα πλασματικό μηδέν, δημιουργώντα μια νέα γραμμή, αυτό δεν είναι πρόβλημα βεβαίω κατά αυτή την έννοια πάντα, και να δείξουμε λοιπόν, να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα στους εταίρου μας, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αφήσει την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, πολιετούς ε, ε, του πολιετούς υπολογισμού χωρίς κανένα περιθώριο, αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, ειδικά εάν συμφωνήσουμε και ακούσουμε προσεκτικά τον πρόεδρό μας που λέει να μην έχουμε διορθωτικό προϋπολογισμό κάθε μήνα. Όμως, είτε έχουμε περιθώριο του 0,1 ή του 0,2 ή κανένα περιθώριο, στην ουσία είναι το ίδιο και το αυτό. Και έχω και ένα καλό νέο για τον σοσιαλιστή συντονιστή. Τι θα γίνει ε, με, το, με τα πιλωτικά προγράμματα στο κεφάλαιο 2 ε, όπου φαίνεται ότι οι πρώτοι υπολογισμοί δείχνουν, έδειχναν τουλάχιστον να υπάρχει ε, έλλειψη ε, μισού εκατομμυρίου. Δεν υπάρχει τέτοια έλλειψη και ελπίζω ότι πραγματικά θα ακολουθήσετε τις προτάσεις μας. Γιατί οι προτάσεις αυτές έγιναν επί, ε, επί συμφωνημένων εκ των προτέρων αρχών. Ε, προσθέτοντας βεβαίως και κάποιες τεχνικές θεωρήσεις οι οποίες δεν αλλάζουν. Εγώ δεν χειραγώγησα τίποτα, εγώ δεν άλλαξα τίποτα, κανέναν αριθμό. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Πρέπει να υπάρχει ένα έγγραφο, το TENRAP έγγραφο, το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχεία τα οποία συζητούμε. Πώς δηλαδή θα δοθούν τα 81 εκατομμύρια για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάκαμψης και επίσης πώς ε, είναι δυνατόν να γίνουν οι 123 ε, πληρωμές για το 2010. Και υπάρχει κι άλλο ένα, ε, κι άλλη μια μπροσούρα που είμαι σίγουρος ότι σας έχει, σας έχει δοθεί που περιέχει όλες τις τροπολογίες οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Συμβούλιο. Είτε τροποποιήθηκαν δηλαδή, είτε απλώς ε, δεν έγιναν δεκτές. Απερίφθησαν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με δύο υποθέσεις. Δηλαδή ότι είτε επανυποβάλλομαι τα πάντα από την πρώτη ανάγνωση και όλα αυτά βρίσκονται στο DOC 10 αλλά ε, στην ουσία θα επικαλυφθεί η ψηφοφορία ε, από την ε, ψηφοφορία του DOC 10 RAP. Δηλαδή, εάν ψηφίσουμε υπέρ της Ίσως θα πρέπει να ψηφίσουμε δηλαδή πρώτα για την επανυποβολή και μετά ε, να ψηφίσουμε για το Doc 10 Rap. Και ελπίζω ότι όλες οι επιθυμίες και όλες οι σκέψεις της ε, Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής ε, θα έχουν βρει την θέση τους στο ψήφισμα ψήφισμα μέσω του οποίου μπορούμε να μεταφέρουμε ο σε τις επιθυμίες και τα μηνύματα της πολιτικής μας ομάδος. Αλλά βεβαίως το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και την ενιαία φωνή μας, την ενιαία φωνή του Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2010. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως ε, την ε, γραμματεία γιατί δούλεψαν πάρα πολύ. Ε, δεν σταμάτησαν ούτε καν το Σαββατοκύριακο έτσι ώστε να έχουμε εμείς αυτή την τελική μορφή όλων των εγγράφων και των τροπολογιών. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τους τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ισηγητά όντως ε, είναι η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μετά από τη συνδιαλλαγή και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή για τον τρόπο με τον οποίο μαζί βεβαίως και με όλη την αντιπροσωπεία ηγήθηκε αυτή της συνδιαλλαγής με την Σουηδική Προεδρία η οποία έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση ε, και για τα πολιτικά προβλήματα αλλά και για τις πολιτικές προτεραιότητες ε, του Συμβουλίου. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε ε, ε, και τον, την Κομισιόν που έπαιξε τον ρόλο του Honest Broker. Από πλευρά Κοινοβουλίου, νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα αυτή τη συνδιαλλαγή. Δεν θα ξαναμπώ σε λεπτομέρειε βεβαίω, αλλά νομίζω ότι τρία σημεία είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να υπογραμμιστούν. Πρώτα λοιπόν πρέπει να βρούμε τον τρόπο να χρηματοδοτήσουμε το σχέδιο ανάκαμψης, recovery plan, και χωρίς καθυστέρηση με βάση τις προθεσμίες που είχαν ορίσει τον, την περασμένη άνοιξη και τα άλλα διαθεσμικά όργανα να ετοιμαστούμε για τη συνδιαλλαγή που χρειάζεται στο 2010. Για το 2009-2010 λοιπόν μπορούμε να βρούμε τα κατάλληλα κονδύλια για τη χρηματοδότηση των δράσεων που έχουν προβλεφθεί από το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης Επενδύσεις ως προς την αναμετατροπή της ενέργειας, ε, στροφή προς, τις, προς καθαρές μορφές δηλαδή, και τις τηλεπικοινωνίες με την ευρυζωνική επικοινωνία, με τον προπολογισμό του 2010. Αφετέρου, όπως είπε και ο Λάσλο, κατά πόσο πιθανότητα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και είναι ίσως και η τελευταία φορά, τουλάχιστον δυνάμει των παλαιών συνθήκων, που δέχθηκε μια πολύ σημαντική δημοσιονομικά τροπολογία αλλά και πολιτικά του Κοινοβουλίου για το γεωργικό προπολογισμό. Έκανε δεκτό το, δεκτή το Συμβούλιο. 300 εκατομμύρια ευρώ, όχι τα 280 που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Ήταν ε, σκληρός διαπραγματευτής ο εισηγητής στο σημείο αυτό. Για τη χρηματοδότηση νέων πολιτικών για την γαλακτοκομική παραγωγή με το λεγόμενο Milk Fund, το Ταμείο για το Γάλα. Επίσης, μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε και στο προγραμματισμό μας και τη χρηματοδότηση για το 2010 των εργασιών για την ε, ενίσχυση ασφάλειας του ε, σταθμού του Κοσλοντούι με μεγάλη επικαιρότητα και σημασία λόγω της συμφωνίας που έχει ασφαλιστεί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και ε, βουλγαρικής κυβέρνησης που δεν είναι δυνατόν ε, να συμπεριληφθεί στην διατύπωση τουλάχιστον την τελευταία στιγμή. Πραγματο... Και από την άλλη έχουμε μια ιδιαίτερη και αναπάντεχη δυσκολία γιατί χρειάστηκαν επιπλέον κονδύλια ε, για τον προϋπολογισμό του 2010. Και εν τέλει η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε τα τρία τέταρτα των απαιτούμενων ε, κονδυλίων που δέχεται υπό τον όρο Fresh Body το Συμβούλιο, δηλαδή χρήματα που προκύπτουν από εξοικονόμηση πόρων υφισταμένων στον ε, γεωργικό προϋπολογισμό, εν μέρη από το μέσο ευελιξίας και κατά ένα τρίτο από τις ε, θυσίες που ε, έκανε εν τέλει που δέχτηκε να κάνει τελικά η προσωπία του Κοινοβούλιο. Φυσικά θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τις ε, δεσμεύσεις αυτές. 81 εκατομμύρια ευρώ ακριβώς θα χρειαστεί να αντληθούν από την κατηγορία 1α. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα, μαζί με τις νέες τροπολογίες που θα μας ε, παρουσιάσει ο εισηγητή μα που τι έχει επεξεργαστεί επί μακρόν με του συντονιστέ. Και συμπληρώνω αυτό που ο Λάσλο, υπενθυμίζοντας ότι αυτή η συμφωνία πρότεινε, πρόβλεπε και την διατύπωση είτε διμερών είτε μερών δηλώσεων το Κοινοβούλιο, τα, θεσμικά, τα άλλα θεσμικά που βλέπετε και στο παράρτημα του σημείου 8 στο έγγραφο εργασίας που έχουμε για τη συνεδρίασή μας, το υπαριθμόν 1. Οι δηλώσεις λοιπόν αυτές, πολύ σημαντικές, η πρώτη είναι πολύ σημαντική ε, νομικά, μια κοινή δήλωση των τριών θεσμικών οργάνων ως προς την συνέχεια της μασονομικής διαδικασίας 2010. Ένα θέμα το οποίο προκαλεί ε, αντιδράσεις εκστατικές από, τους, ε, από πλευράς των ειδικών νομομαθών. Δεν θα τους χαλάσουμε φυσικά τη χαρά και τον ενθουσιασμό. Ένα θέμα το οποίο επανέρχεται. Η δημοσιονομική διαδικασία του 2010 ανεπτύχθη με βραδείς ρυθμούς κατά μια χρονική περίοδο όπου όμως ίσχυε η συνθήκη της νίκαιας. Ολοκληρώνεται όμως τώρα, 1η Δεκεμβρίου, η τελική ψηφοφορία λαμβάνει χώρα στις 16, 17 Δεκεμβρίου, σε χρονική στιγμή καθήν ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Φυσικά από την αρχή προβλέφθηκε η ε, πολιτική συμφωνία φυσικά, αλλά και η ε, επικράτηση της κοινή λογικής, έτσι ώστε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους σε μια λογική διαδικασία με τη συνθήκη της νίκης. Εξευρέθη η νομική εκείνη διατύπωση η οποία επιτρέπει τα ρολόγια να σταματήσουν στις 30 Νοεμβρίου και να χαρακτηριστεί η ψηφοφορία της 17ης Δεκεμβρίου σε μια ψηφοφορία η οποία ελάμβανε χώρα στις 12 παρα λεπτό τα μεσάνυχτα της 30ης Νοεμβρίου. Αυτό είναι για να σας δώσω με μια εικόνα να καταλάβετε τι σημαίνει η κοινή δήλωση υπαριθμών 1. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου που υπογράφει τον προπολογισμό και η υπογραφή του που θέτησε σε ισχύ τον προπολογισμό χρειαζόταν ασφαλώς τις νομικές εγγύησεις, πράγμα το οποίο εξασφαλίστηκε χάρη στη δήλωση αυτή την οποία χρειαζόταν ο πρόεδρος Μπούζεκ για να μπορέσει να υπογράψει. Και Θεωρώ απαραίτητο να αναφέρω επίσης την τροπολογία στο σχέδιο ψηφίσματος του ζήτημου στην οποία πρότεινα ψήφισμα που σχετίζεται με την προφορία στη δεύτερη ανάγνωση με την τροπολογία υπαριθμών 11 της οποίας μόνο στόχος είναι η παραπομπή στην κοινή δήλωση. Έτσι ώστε να πούμε ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει απόψε την κοινή αυτή δήλωση. Τόσο ώστε να διασφαλιστεί ε, πολιτικά ο πρόεδρος Μπούσικ, όσο και για να προστατευτεί η εξαιρετική χαρά των νομομαθών μας. Μετά έχουμε την κοινή δήλωση στο δεύτερο παράρτημα για το ε, θέμα των κτηρίων ακινήτων, πολιτική ακινήτων όλων των θεσμικών οργάνων και των σχετικών υπηρεσιών. Στο υπαριθμό τρία παράρτημα. Επίσης κοινή δήλωση για την απλούστευση και τη διαχείριση διαρθρωτικών μέσων και κονδυλίων συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Υιοθετήθηκε επίσης πολύ σημαντική δήλωση, κοινή δήλωση σχετική με το κεφάλαιο 5, της διοικητικές δηλαδή δαπάνες, η οποία έχει μεγάλη πολιτική σημασία, καθώς επιτρέπει ήδη τη χρηματοδότηση στο βαθμό που υπάρχουν ανάγκες του ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Προέδρου του Συμβουλίου όπως θεσπίζονται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και υπενθυμίζω ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας μετατρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο και δημιουργεί το λειτουργήμα του μόνιμου διαρκώς ε, λειτουργούντος θεσμού του ε, Προέδρου του Συμβουλίου, που είναι σε διαρκή λειτουργία και επαφή με τα άλλα θεσμικά όργανα και που διαφοροποιείται από, τον, ε, από το Συμβούλιο των Υπουργών που έχει πιο έκτακτη μορφή και που χρειάζεται λιγότερα κονδύλια. Μας απευθύνθηκε από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου μια διορθωτική επιστολή για τον προπολογισμό αυτών την τελευταία στιγμή η κατάσταση πολιτικά ήταν ασφαλώς πολύ λεπτή, πολύ ε, ευαίσθητη, διότι προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορούσε να δείξει επιφυλακτικότητα ως προς την, ή μάλλον να εγκρίνει με αίρεση τη χρηματοδότηση του Προέδρου, δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο ήταν εκείνο που πάντοτε διεκδικούσε και υπαστήριζε αυτή τη ε, θεσμική μεταρρύθμιση που προτείνει η Συνθήκη τη Λισαβόνα. και με μεγάλη χαρά βλέπουμε την κατάρριψη των τελευταίων εμποδίων στην κύρωσή της, εξωτερικού αυτή την έκρηξη χαρά και ευδαιμονίας δεν μπορούσαμε να την εκφράσουμε τελικά με επιφυλάξει προ τη χρηματοδότηση για τα είδη χαρτικών ή τα τηλεφωνήματα των υπηρεσιών ε, του Προέδρου του Συμβουλίου. Μεν, αλλά δεν μπορούσαμε δε και να επιτρέψουμε σε ένα θεσμικό όργανο, Συμβούλιο των Υπουργών ή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, να αντλεί από το περιορισμένο αποθεματικό που θα μας περισσέψει το 2010 στον τίτλο 5, που χρηματοδοτεί τις διοικητικές δαπάνες όλων των θεσμικών οργάνων, κονδύλια, ενώ υπάρχει συμφωνία πολιτική μεταξύ όλων των οργάνων, η υιοθέτηση του προπολογισμού του 2010 να λάβει χώρα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι νέες ανάγκες που γεννά η θέση ισχύ της Συνθήκης Λισαβόνας, ανεξαρτήτως της φύσεως ή της προελεύσεως αυτών των ε, αναγκών και είχαμε συμφωνήσει, περιλαμβάνει ακόμη συμφωνία την πρόβλεψη, ότι μόνο με διορθωτικού προπολογισμού θα αντιμετωπιστούν αυτέ οι νέε ανάγκε μέσα στο 2010. Και ξαφνικά το Συμβούλιο αισθάνεται απελπισία και απόγνωση γιατί διαπιστώνει ότι τίθεται σε εφαρμογή συνθήκη τη Λισαβόνα νωρίτερα, πιο, πιο νωρί από ό,τι περιμένανε, δηλαδή το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο του 2010, και σε αυτό δεν είναι έτοιμο και δεν έχει αρκετού πόρου για να λειτουργήσει. Η λύση λοιπόν που βρήκαμε ήταν τέτοια ώστε να εξασφαλίσει ότι το Συμβούλιο των Υπουργών θα χρηματοδοτήσει από τον δικό του προπολογισμό του έτους 2009 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο βαθμό που είναι αναγκαίο και με τα κονδύλια που χρειάζονται για τη λειτουργία του ε, για το 2010 και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Και αυτό γράφεται στο τέταρτο παράρτημα για τον τίτλο 5 ρητά, Αναφέρεται δηλαδή ότι δεν περιορίζεται κατ' ουδένα βαθμό, δεν περιστέλλεται κατ' ουδένα βαθμό με αυτή τη χρηματοδότηση το ε, αποθεματικό του 2010 που θα προβλεφθεί και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των διοικητικών αναγκών όλων των θεσμικών οργάνων και ιδιαιτέρω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα 72 δηλαδή εκατομμύρια ευρώ. Ξέρω ότι μακρηγόρησα στο θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να αντιληφθείτε ότι έχει τεράστια πολιτική σημασία. κρίνουμε άκρως απαραίτητο να βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει προτίμηση από πλευράς του Συμβουλίου ή δικαίωμα εξόνησης για το αποθεματικό αυτό, ότι θα έχει δηλαδή Ε, ότι θα έχει δηλαδή προτίμηση να αντλήσει κονδύλια από το επαθεματικό το Συμβούλιο αυτό θεσμικό όργανο και το Κοινοβούλιο μέσα στη γενεοδορία του υποκλίνεται και χαιρετίζει την εκλογή του κυρίου Φαν Ρόμπο του τα κονδύλια που θα χρειάζεται για τη λειτουργία του ε, θεσμού αυτού το 2010. Για το πέμπτο παράδειγμα τώρα έχουμε να κάνουμε με μια μονομερή δήλωση ή αν θέλετε μπορείτε να τη χαρακτήσετε και δίμερη. Πρόκειται για μια δήλωση τη Επιτροπή, την οποία όμω έχουμε ζητήσει εμεί, για τη μεταγενέστερη χρηματοδότηση του Κοσλοντουή. Γιατί θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί η θέση εκτό λειτουργία και η ασφάλεια του, ε, της μονάδας του Κοσλοντουή. Βρέθηκε λοιπόν μια λύση για το 2010, αλλά παραμένει εκκρεμές το ζήτημα του 2011-2012 2013 που δεν μπορούμε να ε, στηρίξουμε για τη χρηματοδότηση τα αίτια αυτά μόνο στα αποθεματικά. Και γι' αυτό μιλούμε για την δυνατότητα, ανα, όποια στιγμή βρεθεί ε, η δυνατότητα για μια μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση των δημοσιονομικών μέσων, να συμπεριλάβουμε στην αξιολόγηση αυτή, ανάλογα με τις μεσονομικές συμφωνίες που θα ισχύουν, και το Κοσλοντουή. Φυσικά και θα προτιμούσαμε το Συμβούλιο να είχε υποκληθεί στην κοινή λογική και να είχε ανταποκριθεί στις προτάσεις μας. Ε, στο όμως το Συμβούλιο και ως γνωστόν ε, η σιωπή λογίζεται ως συνένεση. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, συμφωνεί να λάβει υπόψη εγώ μάλιστα είχα προτείνει λάβει υπόψη ε, σε πνεύμα ε, σεβασμού, respectfully, ε, που είχα ζητήσει εγώ, το οποίο όμως respectfully κάπου χάθηκε και δεν ξέρω, ίσως για λόγους νομοτεχνικούς, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ μου άρεσε αυτή η λέξη και θα ήθελα να επανέλθει. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι όμω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βρει του απαραίτητου πόρου και θα θυμούνται ασφαλώ οι πιο παλιοί, όπω ο Ράιμερ Μπέγκε ιδιαίτερο, που διαρκώ μα υπενθυμίζει, ότι το πρόβλημα αυτό της διασφάλισης της μονάδα του, του σταθμού του Κοσλοντούι είναι ένα πρόβλημα το οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εσκεμμένος άφησε ανεπίλητο. Πρόκειται για ένα από αυτά τα απολυφάδια, τα leftovers της συμφωνίας 2007-2013 που συνήφθη το 2006 την Άνοιξη, όπου Μιλήσαμε για το Εγκλαλίνα της Λιθουανίας και τον πυρηνικό σταθμό της Σλοβακίας, της οποίας, του οποίου λυσμό το όνομα, Ουρνίτσε. Ε, ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι ο Κοσλόντοϊ θα έπρεπε, γιατί και ε, αυτό είναι ίδιου τύπου σταθμός, ε, άρα θα έπρεπε να επαχθεί στην ίδια διαδικασία κατεργασία και αφοπλισμό, αλλά αφού δεν ήταν ακόμη τότε στην ίδια μοίρα η Βουλγαρία και δεν διαπραγματευόταν με τους ίδιους όρους η κυρία Μιχαήλοβα, η βρετανική κυβέρνηση της εποχής, εργατική και κάπως χερέκακα, γιατί βέβαια αν ήταν άλλη κυβέρνηση θα είχε διαφορετική στάση, η βρετανική στάση εποχή, κυβέρνηση λοιπόν της εποχής είπε «Α, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με κράτος το οποίο δεν ανήκει ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ανέκδοτο φυσικά, γιατί η Βουλγαρία του μεταξύ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι ιδιαίτερω για τη συμμετοχή της ε, στους κόλπους μας, αλλά είμαστε αναγκασμένοι λόγω αυτής της παράβλεψης ε, να βρούμε νέους σπόρους. Εν τέλει, συμφωνήσαμε επίσης και σε μια κοινή διακήρυξη των τριών οργάνων, των τριών θεσμικών οργάνων που χρειάστηκε να κοπιάσουμε για να διατυπώσουμε, για μεταβατικούς κανόνες που ισχύουν ιδιαίτερα ως προς, ε, ως προς τα εμβάσματα και τους διορθωτικούς προϋπολογισμούς που θα επιτρέψουν τη μετάβαση από την Ίκαια στην θήκη της Λισαβόνας, εντολή δηλαδή την οποία ε, μας είχε αναθέσει το, το Κοινοβούλιο, η Ολομέλεια συγκεκριμένα, με βάση είχα παρουσιάσει και με την έκθεσή μου στην Επιτροπή των Προπολογισμών και τη διαπραγμάτευση που οδηγεί σε βελτίωση του αρχικού κειμένου κατά τους όρους που είχαν ζητήσει πολλοί από τους συναδέλφους Τη αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου. Κυρία Κρέσλε, ιδιαίτερος και άλλοι. Και ο Ράιμερ Μπέγκε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κείμενο στο συμπληρωματικό φάκελο, στα Plementary Dossier, υπαριθμόν ένα σελίδα με αναφορά ιδιαίτερα στα άρθρα 22 και 23 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που ρητά αναφέρεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν, εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Είχαμε θεωρήσει ότι είναι αυτονόητο και γι' αυτό δεν το είχαμε σημειώσει ρητά. Πλην όμω οι συνάδελφοι μα επισήμαναν ότι καλό ήταν να σημειωθεί αυτό ρητά ώστε να μην παραμείνει καμιά αμφιβολία. Με το ίδιο πνεύμα διατυπώνουμε σε μια διατύπωση η οποία δεν είναι ακριβώς αυτή την οποία είχε προτιμήσει η κυρία Γκαρσία Σαβά όπου στο τέλος του κειμένου αναφέρει το γεγονός ότι δεν συμφώνησαν ως προς την ε, έγκριση ενό εμβάσματος στα δύο θεσμικά όργανα. Το ένα, μάλιστα, δέχθη το. Μάλλον και τα δύο είχαν δεχθεί την ε, έγκριση ενό εμβάσματος, αλλά σε χαμηλότερα ποσά από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι, κυρία Χαρβάλ, μιλάει για την απλουστευμένη διαδικασία συνδιαλλαγής η οποία μας εκκρίθηκε ότι, ότι δεν ήταν δυνατό ή τουλάχιστον ευχερές να υλοποιηθεί. Και έτσι μπορέσε με τη δήλωση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς να αποσύρει την πρόταση για το έμβασμα, αντί να γίνει ταχυριθμό έμβασμα. Και μετά μπορεί να ξανανοίξει τη διαδικασία, πράγμα το οποίο λίγο πολύ μας φέρει στην ίδια κατάσταση. Μου φαίνεται καλή η συμφωνία, σοβαρή η συμφωνία εξασφαλίζει πιστεύω τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου σε αυτό το μεταβατικό καθεστώς, το οποίο μεταβατικό καθεστώς για το Κοινοβούλιο θα έχει ιδιαίτερη αξία γιατί θα επιτρέψει την θέσπιση μια σειρά κανόνων οι οποίοι για μερικέ εβδομάδε ή μερικού μήνε μόνο μπορεί να ισχύσουν, αλλά ταυτόχρονα θα έχουν και πειραματικό ε, χαρακτήρα. Και εάν αποδειχθούν ε, λογική, αν φέρουν σωστά αποτελέσματα, μπορούμε να τους μονιμοποιήσουμε διαφορετικά, τους ανατρέπουμε και μπορεί να γίνει μια μεγάλη υλοποίηση, μια μεγάλη αναθεώρηση, ευρύτερη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και ε, εν ώψη και της έκθεσης κ. Σίγκεμπορ μπορούμε, μπορούμε να δούμε τα θέματα αυτά. Τελευταία παρατήρηση. Με συγχωρείτε που μακρηγορώ. Έχουν τεράστια σημασία όμως όλα αυτό το θέμα mm. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής των Προπολογισμών ε, τον τρόπο με τον οποίο χειριστήκαμε την εντολή που μας σχεδόσε. Ένα σημείο που έθιξε και ο Λάσλο για το αν επιφυλασσόμεθα με ένα μικρό αποθεματικό στο 1α. Υπάρχει βέβαια. Είναι πειρασμός το να γράψουμε μηδέν πολιτικό μήνυμα του Κοινοβουλίου προς τα άλλα θεσμικά όργανα. Μηδέν ιστοπηλίκων. Εγώ όμως, για λόγους σύνεσης, θα πρότεινα να αφήσουμε ένα μικρό ποσό. Γιατί? Κινδυνεύουμε. Έστω και αν ε, θεωρήσουμε όταν εφείς ε, η άλλη λύση να ε, βρωμίσουμε τα χέρια μας προσπαθώντας να βρούμε μία λύση και ταυτόχρονα να φοβηθούμε με το μηδέν αυτό αποθεματικό να αναπηδήσουμε από χαρά γιατί είναι τόσο χαμηλό το ταβάνι που θα κάνουμε καρούμπαλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι προτιμότερο να έχουμε ένα μικρό αποθεματικό και για τους χρηστές αλλά πάνω απ' όλα για τους υπολογιστές που δεν έχουν τόσο μεγάλη φαντασία όσο οι εισηγητές μας, και όπως πει ο Λάσλο, καλό θα ήταν να μην ξυπνήσουμε μια μέρα για να διαπιστώσουμε την ώρα της ψηφοφορίας, την ώρα που θα κληθεί ο πρόεδρος να θέσει την υπογραφή του στο έγγραφο, του προπολογισμού, ότι το κοινοβούλιο εξαναγκάστηκε να εγκρίνει και ουσιαστικά ο πρόεδρος καλείται να υπογράψει ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα ήταν ε, ασυμβίβαστος, θα ήταν ε, παράτυπος ως προς τη συνθήκη, γιατί ε, λείπουν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Και έτσι θα πρότεινα, μια και είμαστε σε αυτή τη φάση της μετάβαση, να είμαστε πιο επιφυλακτικοί και να διατηρήσουμε ένα μικρό αποθεματικό το οποίο μπορούμε στη συνέχεια να απορροφήσουμε για να χαιρετήσουμε τη μεγάλη μας επιτυχία. Έχουν ζήσει το λόγο οι συγητές και σκιώδεις συγητές. Ε, Χαιρετίζω εδώ την παρουσία του συναδέλφου που <laughs> απεχώρησε ήδη από τη φαίνεται. Χαιρετίζω λοιπόν την απουσία της Αντιπροέδρου κυρίας Ρόδη Κράτσα, η οποία ήταν ε, εδώ πριν και ίσως να γυρίσει πάλι, δεν ξέρω και η οποία από πλευρά του Προεδρείου παρακολουθεί τα θέματα τη ενημέρωση, τη επικοινωνιακή πολιτική και ίσω θελήσει να λάβει το λόγο εφόσον επανέλθει στην αίθουσα και θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή, στους εισηγητές. Ο πρώτος που τον ζήτησε είναι ο Σαλβαδόρ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ ήμουν, ναι, ναι, ήθελα να πάρω το λόγο. Αλλά μετά από το όσο είπε ο Λάσλο και κυρίως μετά από τα δικά σας οφάλα για Πρόεδρε, εγώ τι να πω πια. Τι να πούν και οι συντονιστές οι καημένοι. Μερικά θέματα μόνο επιγραμματικά. Τα εξή τρία. Το πρώτο δεν συνδέεται άμεσα με την τρίτη ανάγνωση, τη δεύτερη ανάγνωση, συγγνώμη, σε ό,τι αφορά τα 25 εκατομμύρια ευρώ ως έξοδα της Προεδρίας του Συμβουλίου θυμίζουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι μια κατεπίγουσα λύση και τίποτα παραπάνω. Διότι χρηματοδοτούμε ε, του 2010 εκ μεταφοράς ε, το 2009. Είναι πολύ σημαντική ε, η συνέπεια αυτή, διότι το, το Συμβούλιο έχει πλεονασματικό προϋπολογισμό. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στις διαπραγματεύσεις του χρόνου για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να παραμείνει το ποσό αυτό. Από το Γενάρη και μετά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα διαπραγμάτευσης με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως επειδή δεν είναι πολύ σαφής η ποσοτικοποίηση. Δεν ξέρω, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει υπολογίσει το τελικό κόστος και τη θέση σε ισχύ και ποιες είναι οι ε, θεσμικές προεκτάσεις ε, τις δημιουργίες της νέας αυτής υπηρεσία και πώς θα επηρεάσει τον προπολογισμό και το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμεί ω Επιτροπή προπολογισμών και ιδιαίτερα ο για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα έχει πολλά να μας πει του επόμενους μήνες, το 2010. Στη συνέχεια, αφορά στο Κοσλοντού η Πρόεδρε, ε, είναι ακριβής. Τελικά, η συμφωνία δείχνει ότι η διαπραγματευτική ομάδα που στείλαμε στη συνδιαλλαγή έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Διότι μπήκαμε λέγοντα ότι το Κοσλοντόι δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί εις βάρος της κατηγορίας 1 και τελικά βγήκαμε από τη συμφωνία και τη συνδιαλλαγή ακριβώς με ε, αυτή τη νίκη. Δηλαδή με φρέσκο χρήμα και όχι αναδιάταξη πόρων από αλλού. Ήταν πολύ ισχυρή η θέση μας και μπορεί να σόκαρε τους Βουλγάρους ε, φίλους μας ε, στην αρχή, αλλά αυτό το επιτάσσει η δημοσιονομική λογική. Αυτό που δεν γράφει ο προπολογισμό, το προσχέδιο προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου δύσκολα μπορεί να μπει στη συνδιαλλαγή. Βρέθηκε η μόνη δυνατή λύση δηλαδή που είναι να βρει φρέσκο χρήμα, fresh money το λένε αυτό το Συμβούλιο και να βάλει το χέρι στην τσέπη. Αυτό είναι καλύτερη λύση για όλους και θα το χαρακτήσω και από τα βασικότερα επιτεύγματα άλλωστε της ιδιαλλαγής. Για όλα τα υπόλοιπα που λέει ο εισηγητής ο κύριος Σούριαν, ως ομάδα συμφωνώ απολύτως εγώ και ε, για την πολιτική συνοχή. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε σπιθαμή πίσω, διότι το μήνυμα που θα στέλναμε σε όλες αυτές τις χώρες που ισχυρά εξαρτώνται από την ε, ε, πολιτική συνοχή θα ήταν πολύ λανθασμένο. Τελικά λοιπόν για τις πληρωμές εθετήσαμε ένα ποσοστό πάρα πολύ ε, καλό για το Κοινοβούλιο και μπορεί να το δεχτεί και είναι απορία άξιων που σταμάτησε το Συμβούλιο της διαπραγματεύσεις στο ποσοστό αυτό. Μοιράζει, πολύ ωραία είναι και πολύ καλά τα πήγαμε. Αυτά. Για ένα τρίτο τελευταίο πρόεδρε. Για το μικρό υπόλοιπο της κατηγορίας 1α, ε, το πλεόνασμα, το είπαμε και στην προπαρασκευαστική συνεδρίαση και το είπα και εγώ στο Σούριαν. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να απορροφήσουμε απολύτως το περιθώριο αυτό για λόγους στρατηγικούς. Ε, δεν θα πρέπει να το αφήσουμε με μηδενικό υπόλοιπο. Δεν είναι το ίδιο και το γνωρίζουν όσοι παλιές εδώ καραβάνες στις διαπραγματεύσεις του προπολογισμού. Δεν είναι το ίδιο στην πρώτη ανάγνωση και στη δεύτερη να αφήσουμε με μηδενικό υπόλοιπο το αποθυματικό. Και εδώ απευθύνομαι κυρίως στον συνάδελφό μου Γιώραν Φάρμ. Η πολιτική ανάγνωση έχει σημασία. Είναι άλλο να αφήσει σε πρώτη ανάγνωση μηδενικό αποθεματικό και άλλο σε δεύτερη. Ανοίγει δυνατότητα, ένα παραθυράκι για τη συνδιαλλαγή. Τώρα έχουμε μαθηματικό υπόλοιπο σε δεύτερη ανάγνωση μηδέν, είναι αν μη τι άλλο ρήψο κίνδυνο και δίνει και ένα λάθος μήνυμα. Ότι ψηφίζουμε περιθώρια απλώ για λόγου στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή απόφαση τη Επιτροπή Προπολογισμών. Μπορεί αυτό να είναι λόγο ύπαρξη άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών εδώ μέσα που είναι επιτροπές που πανούν, αλλά ποτέ η Επιτροπή Προπολογισμού που έχει ως στόχο να βάλει μια τάξη και μια, ένα εξορθολογισμό και κυρίως στη δεύτερη ανάγνωση μεταξύ ε, εσόδων και εξόδων. Το σημαντικότερο λοιπόν και το, ίσως και για λόγους τύπου και για λόγους ουσίας καλό θα ήταν να αφήσουμε άθικτο το αποθεματικό 0,7 εκατομμύρια ευρώ, να μην τα πειράξουμε αυτά, να τα αφήσουμε εκεί που είναι και να μην βαθύνουμε περισσότερο γιατί μπορεί να έχουμε έτσι, μαθηματικό, λογιστικό κίνδυνο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Ευχαριστώ πολύ, Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ βεβαίως θα, ήθελα να συγχαρώ τον ε, Σούριαν καθώς επίσης και τον ε, Πρόεδρο για, για, το, για την έκβαση, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Γιατί νομίζω ότι παρέμειναν όλες οι προτεραιότητες ε, άφικτες και επίσης όλοι έδειξαν πολύ καλή διαγωγή όσον αφορά την εξέβρεση των 81 εκατομμυρίων. τα διαφορά με την πρώτη ανάγνωση. Και εγώ ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι δεν θα πρέπει να κατεβούμε παρακάτω από τα στοιχεία της Επιτροπής και γενικώ αυτό είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα σωστής, ορθής ανάλυσης των αναγκών ε, σωστής ιεράρχησης των προτεραιοτήτων ε, και των περιθωρίων. Και νομίζω ότι ήταν καλό βέβαια ότι και μεταξύ των πολιτικών ομάδων υπήρξε ένα πνεύμα συμφωνίας και επομένως εδώ είχαμε μια καλή διαδικασία. Επίσης, είναι γεγονός ότι με τον Γιώραν Φεν είχα συμφωνήσει ε, και προτείναμε κάποια επιπλέον ε, κονδύλια για την ε, δημοσιονομική εποπτεία. Βεβαίω είναι μια πολύ μικρή γραμμή του προπολογισμού. Παρόλα αυτά, αν κατάλαβα καλά, θα υπάρξει παρόλα αυτά ένα μικρό υπόλοιπο και ας το αφήσουμε έτσι όπως είναι. και νομίζω ότι αυτό το μηδενικό υπόλοιπο δεν είναι αυτός σκοπός, δεν είναι στόχος μας. Επίσης νομίζω ότι είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά το πλαίσιο συνεργασίας ε, στην, στις δηλώσεις ε, όσον αφορά και την μετάβαση από την παλιά στην νέα συνθήκη και νομίζω ότι το αποτέλεσμα γενικά ήταν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, η έκβαση πολύ ορθή και χαιρόμαστε. Σχετικά ε, με τις ε, ερωτήσεις του Σούριαν για το πώς θα οργανώσουμε ε, την ψηφοφορία. Ο Σούριαν θα αποφασίσει μαζί με, τους, μαζί με τον Πρόεδρο. Το αφήνω σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Άννα, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα επίσης να πω στην Άννα ότι λυπούμεθα που η συνδιαλλαγή αυτή έγινε τη απουσία της, αλλά βεβαίως ε, ε, εκπροσωπήθηκε αποτελεσματικότατα αλλά νομίζω ότι η συμφωνία έγινε πολύ γρήγορα πριν προλάβει να έρθει η Άννα. Και αυτό διότι το Συμβούλιο άλλαξε την τελευταία στιγμή την ε, ημερομηνία, την έβαλε 24 ώρες πριν πράγμα που δυσκόλεψε λίγο τη, κάποιους συναδέλφους, μεταξύ των οποίων και η Άννα. Δράτω με τις ευκαιρίες, μια και αναφερόμαστε σε προσωπικά προβλήματα, για να πω ότι η Γιούτα Χάου δεν είναι ο εξεβονίμων μου, διότι είχε μια δέσμευση, μια άλλη συνεδρίαση που είναι η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση ΑΚΕ. Άρα δεν θα συμμετάσχει σήμερα το απόγευμα στις εργασίες μας. Και αυτό που είναι πιο ε, ενοχλητικό είναι ότι το σύνολο των πρασίνων δεν μπορεί να παρίσταται, γιατί έχουν συνεδρίαση της ομάδας τους εκτός Βρυξελών, σε ένα εξωτικό μέρος, το οποίο φαίνεται ότι απειλείται ιδιαίτερος από την υπερθέρμανση του πλανήτη και που δυστυχώς δεν τους δίνει την δυνατότητα να βρίσκονται εδώ έτσι ώστε να τους δείξουμε πόσο τους αγαπούμε. Λέει ο Πρόεδρος. Συμμετέχουν προφανώς στην συνένεση, αλλά ε, δεν ε, έχουμε εκπρόσωπό τους παρόντα. Όμως, η σοσιαλιστική ομάδα είναι εδώ, ε, εκπροσωπείται με μεγάλη ρόμη και ο Γιώραν ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος και θα ασχοληθώ μόνο με τα υπολείποντα ε, προβλήματα, γιατί νομίζω ότι η γενική αξιολόγηση όσον αφορά την έκβαση της συναλλαγής ε, είναι σαφής. Προστασία των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, πράγμα που έγινε. Ε, συγχαρητήρια στον Λάσλο, γιατί κινήθηκε πάρα πολύ σωστά ακολούθησε την με πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και πραγματικά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γι' αυτό. Πρώτον, γενικά σχόλια. Χαίρομαι που στην συνεδρίαση των συντονιστών την προηγούμενη εβδομάδα καταφέραμε να έχουμε συνένεση σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων των σχετικών με τα 81 ε, εκατομμύρια που θα έπρεπε να ε, δοθούν στις προπαρασκευαστικές δράσεις καθώς επίσης ε, και εις την διευκόλυνση της μικροπίστοσης τα υπόλοιπα όντως χρήματα ε, να μπουν σε διάφορες προτεραιότητες και όχι σε μία γραμμή και μόνο. Όμως, όσον αφορά ε, τις ε, μικροπιστώσεις, έστω και αν φτάσουμε σε συμφωνία στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, ε, όπου είπαμε ότι θα δοθούν 25 εκατομμύρια από το φρέσκο χρήμα. Αυτό όμως αποτελεί ακόμα ε, ε, αντικείμενο διαπραγμάτευση μεταξύ του εισηγητού της Επιτροπής Απασχόλησης και την Επιτροπή. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα πρέπει ο συντονιστής μας, ο, συγγνώμη, ο εισηγητής μας να συμμετάσχει σε αυτόν τον τριμερή διάλογο που θα πρέπει να υπάρξει ή τέλος πάντων να στείλει ένα μήνυμα ε, ε, έτσι ώστε να λυθούν τα προβλήματα τα οποία φαίνεται να υπάρχουν, τουλάχιστον υπήρχαν μέχρι πριν από μια εβδομάδα, μεταξύ της Επιτροπής και της ε, Επιτροπής Απασχόλησης. Ένα σχόλιο τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα για τα στοιχεία του προϋπολογισμού και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην συζήτηση για την γραμμή των δημοσιονομικών υπηρεσιών. Βασιζόμαστε σε μία ίδια εγκριθήσα έκθεση. Ε, είχαμε υποβολή τροπολογιών από την ε, Οικονομική Επιτροπή. Και βεβαίως ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τις 700.000 αντί τις 140 ε, που είχε ζητήσει ο ε, εισηγητής ε, και φαντάζομαι ότι εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η πρόταση η οποία φαίνεται ότι βρίσκει σύμφωνους και τους φιλελεύθερους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να φτάσουμε στις 700.000. Εάν μετά από αυτό εξακολουθεί να υπάρχει υπόλοιπο στην, να υπάρχει υπόλοιπο στην κατηγορία 1α, φαντάζομαι ένα μικρό υπόλοιπο, Μπορούμε να κάνουμε βέβαια μια φιλοσοφική συζήτηση σχετικά με το εάν ε, θα πρέπει να έχουμε μηδενικό υπόλοιπο ή 100.000 υπόλοιπο ή κάτι τέτοιο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το να αφήσουμε ένα υπόλοιπο όμως υπάρχουν και άλλα κεφάλαια ε, στα οποία έχουμε μηδέν. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει σε μερικές περιπτώσεις να βάζουμε υπόλοιπο μηδέν. Αλλά αυτό είναι μια φιλοσοφική συζήτηση η οποία δεν με αγγίζει. Δεν έχουμε, εγώ δεν έχω πρόβλημα εάν κρατήσουμε κάποιο υπόλοιπο με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρεθούν τα χρήματα τις 700.000 που ανέφερα προηγουμένως. Επίσης κάποια άλλα σχόλια. Πολύς λόγος έγινε για την ε, ε, στρατηγική επικοινωνίας ε, και όσον αφορά και για το υπόλοιπο και το, το υπόλοιπο αποθεματικό μάλλον όσον αφορά τις δράσεις επικοινωνίας. Ε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ακολουθήσουμε και εδώ την πρόταση ε, του εισηγητού μας που ταυτίζεται και με τις προτάσεις που μας έδωσε η υπηρεσία, η διεύθυνση μάλλον επικοινωνίας του Κοινοβουλίου. Ένα τελευταίο μικρό σχόλιο. Έχουμε και άλλη μια επιφύλαξη στο Other Management Expenditure, λοιπές δαπάνες όσον αφορά αυτό το αποθεματικό στις λοιπές δαπάνες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βασιστούμε στη νομική βάση της Όλαφ. Ε, νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι όχι απλώς να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα διάφορα αποθεματικά, αλλά όταν θα έχουμε ε, την ε, απάντηση που θέλουμε να αναλάβουμε τις ε, δεσμεύσεις, να προχωρήσουμε με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Ε, γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως το αποθυματικό μπορεί να δοθεί ε, σε μελέτες, αλλά σίγουρα χωρίς να ξεπερνάμε τα όσα έχουμε αποφασίσει για την Όλαφ. Νομίζω και εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια χωριστή ψηφοφορία. Επίσης θα επανυποβάλλω με κάποιες από τις τροπολογίες πάντα ευθυγραμμισμένες με την πρώτη ανάγνωση όμως μπορούμε και οφείλουμε να συμφωνήσουμε με τα περισσότερα από τα στοιχεία. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώραν. Ε, ε, ε, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής ιδιαίτερα στον τρόπο με τον οποίο ο Γιώραν Φέρμ καθ' όλη τη διάρκεια του δύσκολου αυτού εγχειρήματο της διαλλαγή μας, βοήθησε να καταλήξουμε στο τελικό συμβασμό. ε, βεβαίως υπερασπιζόταν πάντα τη θέση τη ομάδα του, αλλά με πνεύμα επικοδομητικό. Και μας βοήθησε και ε, λόγω της γνώσης του της ουηδική γλώσσας σε κρίσιμες στιγμές. Ο Βλάντιμιρ Μάνκα ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς. Πολύ ε, θετικά αυτά που είπατε. Ακόμα και αν έχουμε δύο εισηγητές, καμιά φορά τα πράγματα μπορούν να πηγαίνουν πολύ καλά. Μερικά σχόλια και παρατηρήσεις. Ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει λήξει. Έχει διεκπαιρεωθεί και ολοκληρωθεί σε πρώτη ανάγνωση. Οπότε δεν χρειάστηκαν και προσαρμογές ε, προϋπολογισμούς άλλων πολιτικών ομάδων. Για τα λοιπά λοιπόν ε, όργανα, τα λοιπά τμήματα, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι τα μέτρα που λάβαμε σε πρώτη ανάγνωση για τον προπολογισμό των άλλων ε, οργάνων οδηγούν σε εξοικονομήσεις ε, χρημάτων που μπορούμε να δώσουμε στο σχέδιο ανάκαμψης. Στις μεταφορές πιστώσεων δηλαδή έχουμε μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης και βελτίωσης των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ελπίζουμε τώρα και στην κτηριακή πολιτική να βρούμε τη σωστή πολιτική. Πριν τη συνεδρίαση της συνδιαλλαγής χρειάστηκε να εκδοθεί κοινή δήλωση του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κτίρια. Συμφωνώ πάρα πολύ με αυτή τη δήλωση. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες των κτίριων, είναι πολύ σημαντικό τμήμα των διοικητικών ε, δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μια στρατηγική μέσο πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη με διαπραγματεύσεις. Γνωρίζουμε ότι λύγει σύντομα το δημοσιονομικό πλαίσιο και προσπαθήσαμε να εκπονήσουν και να προετοιμάσουν στρατηγική όλα τα θεσμικά όργανα. Και δεν έχει νόημα, δεν αρκεί το κάθε όργανο να έχει τη δική του ξεχωριστή κτηριακή στρατηγική, αλλά χρειάζεται και εδώ συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων για να μπορούν να εξοικονομηθούν πολυ πολύ πολύ τιμή πόρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Α, συγγνώμη, ένα τελευταίο σχόλιο που ξέχασα. Συχνά παρατηρείται το εξή. Υπάρχουν μέθοδοι χρηματοδότησης των κτηρίων που ε, κάνουν το κόστος να εκτοξεύεται τελικά. Ελπίζω σύντομα να μας προτείνει εναλλακτικέ λύσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Σεγητά. Κυρία Τζεντρεύσκα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου και εγώ να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τον Πρόεδρο που έκαναν τόσο καλή δουλειά. Είμαστε νομίζω όλοι πολύ ευχαριστημένοι, πολύ ικανοποιημένοι από την δεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, Ίσως θα έπρεπε να μιλήσουμε για ε, αριστοτεχνικό προϋπολογισμό, για μαγική θα έλεγα ε, διαμόρφωση, ταχυδακτηλουργική διαμόρφωση του προϋπολογισμού. Πώς φτάσαμε σε αυτό το πέμπτο κεφάλαιο, πώς φτάσαμε να έχουμε αρκετά κονδύλια μέσα από την κατηγορία 5. Ας μην βιαστούμε όμως να ζητοκραγαβάσουμε. Δεν τα έχουμε ακόμα στα χέρια μας τα χρήματα αυτά. 80 με 90 εκατομμύρια ευρώ θα χρειάζονταν για τις ε, ανάγκες μας ε, προσωπικό. στο κεφάλαιο, στο τίτλο 5 υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και ενδέχεται του χρόνου να μην πετύχει πάλι ταχυδακτηλουργία. Να μην ξαναζήσουμε το ίδιο θαύμα. Και πια θα έχουμε ήδη τη συνθήκη της Λισαβόνα σε ισχύ και καμιά ειδική μεταχείριση. Η κατηγορία 5 λοιπόν εγώ θα προτιμούσα να έχει επαρκή πρικοδότηση ώστε να ε, πληρώνει τις ε, δεσμεύσεις της χωρίς δυσκολίες. Ευχαριστώ κύριος Βούγγεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βούγγεν όπως και οι λοιποί συνάδελφοι καλώς ορίζω και εγώ τις εξελίξεις και την έκβαση αυτών των συζητήσεων με την ε, επάνωδο στο προσχέδιο του προϋπολογισμού Νομίζω ότι έχουμε βρει μια καλή λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε, αν και πάντοτε υπάρχουν δυσκολίες, όπως όλοι γνωρίζουν. Δεν υπάρχουν αθευματουργές λύσεις. Επίσης ε, κάποια από τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί όσον αφορά το μέλλον. Κάποιοι συνάδελφοι παραδείγματι αναφέρθηκαν στο γεγονό ότι είναι πολύ μικρά τα αποθεματικά και έτσι ότι στο μέλλον να είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι προτεραιότητες που θα θέλαμε. Η τελευταία συνάδελφο μίλησε για ζητήματα προσωπικού και χρηματοδότηση από τον τίτλο υπαριθμών 5 που θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον, όπως το κλείσιμο του σταθμού του Κοσλοντούι. Εν γέννη πάντως θεωρώ ευπρόσδεκτες αυτές τις ε, εξελίξεις. Ιδιαίτερα όμως, Πρόεδρε, θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή της παρέμβασής σας, τις ε, συμπληρωματικές δηλώσεις, ιδιαίτερα αυτή που αφορά ε, τη συνοχή, την πολιτική της συνοχής και τη χρηματοδότησή της. Τη διάβασα με μεγάλη προσοχή, είναι πολύ επιτυχη η διατύπωση και πιστεύω ότι θα την υποστηρίξουν τη δήλωση αυτή όλοι οι συναδελφοί. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και να υλοποιηθεί. Γιατί αν δεν υπάρχει ικανοποιητικό μηχανισμό σε θέση λειτουργία τη ε, πολιτική συνοχή, ε, αν δεν υπάρχει δυνατότητα να επιταχύνουμε τι δράσει μα με, με την κατάλληλη χρηματοδότηση, θα μείνουν όλα αυτά ωραία λόγια, αλλά χωρί αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και είμαι βέβαιο ότι συμμερίζεται την άποψή σα και ο επόμενο ομιλητή, James, ομιλητής James Ellis. Δεν είμαι βέβαιος, λέει στα γαλλικά ο κύριος Έλλης. Μια που μιλάτε τόσο λαμπρά τη γλώσσα μου, το ανταποδίδω και μιλώ τη δική σας. Θα ήθελα να θέσω τα εξή τρία ζητήματα. Πρώτον, στο παράρτημα 4, την κοινή δήλωση του τίτλου 5, λέγεται στα αγγλικά και επανέρχομαι στη μητρική μου, ότι η προτεραιότητα χρήσης του περιθωρίου στο τίτλο 5 θα πρέπει να δοθεί σε επιπλέον χρηματοδότηση ε, των συνεπειών της θέσης σε ισχύ της συνθήκης της Αβώνας. Υπάρχουν υπολογισμοί, ήδη έχει κάνει υπολογισμούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, τώρα που έχει αρχίσει να ισχύει, όπως λέτε πολύ, ε, σωστά. Γιατί θα μας εξέπλησε αν δεν είχε κάνει τους υπολογισμούς της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το τι κοστίζει η συνθήκη της Λαβόνα ή πώς αλλάζουν οι δαπάνες και τα έξοδα. Ένα δεύτερο τώρα σχόλιο. Κοιτώντα το ψήφισμα που θέτει πλέον σε ισχύ και υλοποιεί το παράρτημα 4, οι συγκεκριμένες παραγράφους 34 και επόμενες 35-36 λέγουμε ότι θα πρέπει να γίνει ε, σε βάθος ανάλυση και ε, αξιολόγηση των δαπανών για περαιτέρω και μελλοντική εξοικονόμηση. Δεν θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τη γραμματεία μας να ψάξει ήδη πού μπορούμε να βρούμε κάποιες δαπάνες, δηλαδή στις 30 Απριλίου κάποια χρονική στιγμή να κάνουμε μια συλλογική παρουσίαση για να έχουμε μια ιδέα που μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα μας χρειάζονται κάποια κονδύλια. Ιδιαίτερα στη χώρα μου και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης Βλέπουμε δημοτικά συμβούλια ή φορείς τοπικής αυτοδιοίκηση που παγώνουν μισθούς ή απολύουν εργαζομένους ακριβώς για λόγους ταμιακούς, διότι το ταμείο τους έχει στερέψει. και αν δούμε ότι αυξάνεται το μισθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση 3,5% ε, δεν είναι καλή εντύπωση και δείχνει ότι η δημοσιονομική αρχή δεν έχει κάνει τη δουλειά της καλά. Να κοιτάξουμε λοιπόν αν μπορούμε στη δίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να κάνουμε οικονομίες. Δεν προτείνω ε, πάγωμα των μισθών ή πάγωμα των επιδομάτων των οικογενειακών ή των τέκνων, γιατί θα εκραγεί το σύμπαν, ε, αλλά να κοιτάξουμε λίγο πώς μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Να το ψάξουν λοιπόν οι Γενικοί Γραμματείς των Θεσμικών Οργάνων. Θα ήταν και αυτή μια ιδέα. Ένα τελευταίο στοιχείο και επανέρχομαι στη γλώσσα μου γιατί είναι πιο τεχνικό. Στο έγγραφο του Ράιμερ Μπέγκε για την κινητοποίηση όχι ακριβώς, πώς το λέμε αυτό, την ενδιάμεση αναθεώρηση και πώς θα χειριστούμε ε, όλα αυτά τα μέσα. Αυτό που λέγει στο τέλος του κειμένου του είναι ότι θα ήθελε τα θέματα αυτά να συμπεριληφθούν και στην ακρόαση όταν γίνει. Εντάξει, είναι λίγο ημομηξία να κάνουμε ακρόαση με δικό μα συνάδελφο, αλλά επειδή είναι δύσκολα τα θέματα και καθόλου. Δεν ξέρω ποια είναι η ημερομηνία. ίσω τη δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου, ωστότε δεν θα ξανασυνεδριάσει η Επιτροπή Προπολογισμού. Πότε θα το συζητήσουμε αυτό, θα μα δώσει η Γραμματεία ένα ερωτηματολόγιο, ε, κάποια θέματα να προετοιμάσουμε για την ακρόαση. Γιατί πολλοί δεν θα ε, γυρίσουμε μέχρι τις 11 Ιανουαρίου και θα έχουμε αμέσως μπροστά μας την ακρόαση. Μια συζήτηση και απουσία ενδεχομένω στο δημοσιογράφο να δούμε τι θέλουμε να το ρωτήσουμε. Merci, Je vais vous répondre sur ce point. Ευχαριστώ αγαπητέ συνάδελφοι. τελευταία Ingeborg Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ζήτησα το λόγο αφού μίλησε ο Γιώραν Φάρμ για το Όλαφ, εντάξει καλά έκανε, ευχαριστώ πολύ, γιατί είναι άλλη το πρόβλημα και θα πρέπει να παίξει ρόλο στι αγροάσεις των υποψηφίων επιτρόπων. Γιατί ήδη παρακάμπτουν, εξαιρούν ε, το θέμα της καταπολέμησης της απάτης και πραγματικά είναι ε, κάτι ε, για το οποίο ανησυχούμε. Τώρα, για τις μελέτες παρακαλώ να διατηρήσουμε το αποθεματικό. Να σας πω γιατί μπορεί να έχουμε τις οργανώσεις που πήραν τα χρήματα, αλλά δεν ξέρουμε τι τα κάνουνε. Ας πούμε εδώ λέει Lloyd, πέντε φορές. Δέκα εκατομμύρια συνολικά ευρώ. Και πού πήγαν, τι, τι θέλουμε τη Λόιτ και με τόσα λεφτά και τι κάνει, τι μελέτες κάνει. Η Deloitte η Oceanic Development SAS. Ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν κάτι εκατομμυριάκια και αυτοί, τι τα κάνουνε, τι μελέτες έχουμε παραγγείλει εκεί, ποια θέματα διαπραγματεύονται. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι κάτι το εφικτό να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια σχόλια από πλευράς μου. πριν μας απαντήσει και ο εισηγητής και πριν εξάγει τα τελικά του συμπεράσματα. Σχετικά με την παρατήρηση του Σαλβαδόρ Καρίγκα. Θα ήθελα να πω στην Επιτροπή Προϋπολογισμών ότι ο πρόεδρος Μπούζεκ ήρθε την προηγούμενη εβδομάδα πρώτα στην ετήσια συνάντηση, συνεδρίαση των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και μετά το ίδιο βράδυ οργάνωσε δείπνο εργασίας με τους ε, Προέδρους των 6 ή 7 επιτροπών ε, που ε, της αφορά αυτό το θέμα των εξωτερικών μελετών. Αύκο, νομική, προϋπολογισμοί, έλεγχος προϋπολογισμού διεθνές εμπόριο και ανάπτυξη. Αυτές είναι, 7 νομίζω ήταν αυτές οι επιτροπές. Διαπιστώσαμε λοιπόν πρώτον ότι έπρεπε το Κοινοβούλιο επιγόντως να συστήσει ομάδα εργασίας Task Force συνεργασίας με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να δουλέψουν επί της ε, προτάσεως ε, του καταστατικού αυτής ε, της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Επίσης, κυρίως διότι το Συμβούλιο ήθελε να έχει ολοκληρώσει μέχρι τον Απρίλιο όλη τη διαδικασία με τις αποφάσεις και τα λοιπά. και βεβαίως υπεύθυνη θα ήταν ε, για το θέμα αυτό η κυρία Άστον. η οποία θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία στη διάθεσή της ε, μέχρι τον Απρίλιο, μέχρι τέλη Απριλίου. Υπήρξε λοιπόν ζήμωσης ανάμεσα ε, στις στις δύο επιτροπές οι οποίες διεκδικούσαν την προεδρία αυτής της ε, Task Force. Τελικά μάλλον ε, αποφασίστηκε ότι η ΑΦΕΤ θα ήταν ε, υπεύθυνη, αλλά οπωσδήποτε σε αυτήν την Task Force θα υπήρχαν εκπρόσωποι όλων των αρμοδίων κοινοβουλευτικών επιτροπών και επομένως οπωσδήποτε θα υπάρξει εκπρόσωπος και στις επιτροπές Προϋπολογισμών. Και όταν θα υπάρξει πλέον πολιτική συμφωνία, τότε θα μελετηθούν υπεραιτέρω ε, λεπτομέρειες, νομικές ε, κλπ. Όσον αφορά τις ε, παρατηρήσεις του Γιώραν Φεν, λαμβάνω υπόψη την πρόταση που έκανε να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή απασχόλησης έτσι ώστε να προετοιμαστεί ο τριμερής διάλογο ο οποίος θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα και επομένως ναι θα έρθουμε σε επαφή με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Επίσης να πω ότι έχετε στα έγγραφά σας μια επιστολή της κυρίας Ντόρις Πάκ ε, Προέδρου της Επιτροπής ε, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης, ε, ε, βάσει της οποίας έρεται η επιφύλαξη της Επιτροπής αυτής. Όμως, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικής αρχής όσον αφορά το υπόλοιπο μηδέν και το να γράψουμε υπόλοιπο μηδέν και έπειτα, από την άλλη πλευρά, υπάρχουν πρακτικά προβλήματα. Εγώ, σαν Πρόεδρο, πρέπει να επιστήσω την προσοχή σα στα, πρακτικά προβλήματα. Θα πρέπει, επομένω, να βρούμε λύση στο να υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση όλων των ε, χρηματοδοτικών και δημοσιονομικών εργαλείων που θα εφαρμοστούν του χρόνου και η γραμματεία μου λέει κατά αυτή την έννοια ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το υπόλοιπο της κατηγορίας 5. και ενώ στην αρχή μιλούσαμε για 72 εκατομμύρια, ε, τώρα καταλήγουμε στα 74, κάτι εκατομμύρια. Ε, όμως στην κατηγορία 1α εξακολουθούν να λείπουν περίπου 200.000 ευρώ ε, βεβαίως από πολιτικής απόψεως ε, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα υπόλοιπο το οποίο είναι σχεδόν μηδενικό. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να δούμε εάν μας συμφέρει κατά κάποιο τρόπο απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα να έχουμε αυτό το, το, το υπόλοιπο μηδέν. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μεσάνυχτα βάλαμε ε, ε, τα κοντέρ πάλι στο μηδέν και επομένως θα πρέπει να δούμε εάν και κατά πόσο θα αλλάξει και η τακτική του ε, Συμβουλίου. Ξέρουμε ποια είναι τα πλαφόν, ξέρουμε ποια είναι τα κατόφλια, από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί και η Επιτροπή και το Συμβούλιο. Όσον αφορά το ερώτημα που έθεσε ο James Ellis για την ακρόαση μαζί με τους συντονιστές καταλήξαμε στην εξή λύση. Δηλαδή, να ακολουθήσουμε τις γραπτές ερωτήσεις, που δεν ξέρω ποιος έχει συγγράψει το έγγραφο αυτό, ποιος έχει εκπονήσει, δεν ξέρω ποιο το εκπώνησε το έγγραφο αυτό. Πάντως έχουμε καταλήξει σε κάποιες ερωτήσεις γραπτές οι οποίες ε, είναι ανόητε οι οποίες όμως κατά κάποιο τρόπο είναι κοινέ για όλες τις επιτροπές και φαίνεται ότι αντιπροσωπεύουν μια κοινή αξία και ένα κοινό βάρος ας πούμε για όλες τις επιτροπές και επομένως να εκτυπήσουμε τις απαντήσεις στις ίδιες ερωτήσεις. Νομίζω ότι στις ε, γραπτές <laughs> στις γραπτές ερωτήσεις θα έχουμε γραπτές απαντήσεις, όπως λέμε στη Γαλλία λέει ο Πρόεδρος, στις κουτές ερωτήσεις έχουμε κουτές απαντήσεις κατά τα λοιπά, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη και την προσωπικότητα ε, του, ε, του υποψηφίου, ε, να έχουμε μια διαδικασία catch the eye, όποιος σηκώσει το χέρι του να πάρει το λόγο. Βεβαίως να, θε, να τεθούν ερωτήσεις ε, επί της πολιτικής που έχει ακολουθήσει ο υποψήφιος και οποιασδήποτε άλλες τέλος πάντων ερωτήσεις ε, οι συντονιστές θα έχουν ε, θεωρήσει σκόπιμες. Νομίζω ότι είναι παράλογο, κυρίως με αυτόν τον υποψήφιο, να ακολουθήσουμε διαφορετική ή ιδιαίτερα τυπική διαδικασία. Πάντως, σε γενικές γραμμές ε, ε, λέμε ακρόαση, η οποία δεν θα ξεπερνάει ε, τα, τις τρεις ώρες. Και να ξεκινήσει η ακρόαση αυτή με προφορική παρουσίαση του υποψηφίου 10 ή 15 λεπτή για να υπάρχει πολύ χρόνος και χώρος για ανταλλαγή απόψεων, ρωτήσεων κτλ. Στρέφομαι τώρα προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Γενικός Διευθυντής επιθυμεί να απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν κυρίως όσον αφορά την αξιολόγηση πιστώσεων ε, για μελέτες ε, ή όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες, κυρίως στα πλαίσια της υλοποίησης και εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας κτλ. ή επί κάποιου άλλου θέματος Θέλετε να πάρετε το λόγο κύριε Γενική Γραμματεύ, α, ε, κύριε Γενική Διευθυντά, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχάς επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με τα λόγια σας ε, για να ορτάσουμε τη σημερινή ημέρα της 1 η Δεκεμβρίου. Σε ό,τι αφορά ε, τα ζητήματα και τις ερωτήσεις που έκανε ο James Ellis για την εξωτερική υπηρεσία. Βεβαίως, και προφανέστατα οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν εργαστεί σκληρά και σύντομα θα έρθουν οι ε, προτάσεις, αλλά από τον ύπατο εκπρόσωπο, ξέρετε, που, την ύπατη μάλλον, ε, που θα κάνει τις προτάσεις της μετά από έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, οι ε, δημοσιονομικές δημοσιονομικέ συνέπειε τη αίσθηση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα σε διοικητικό επίπεδο πάντα, αν υπάρξουν, θα αφορούν ε, την ανάγκη ε, πρόσληψης εθνικών διπλωματών που έχουν κάπως διαφορετικό καθεστώς ε, και ως προς το κόστος τους. Οι προτάσεις όμως αυτές θα φτάσουν από την ύπατη εκπρόσωπο που είναι και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό ως προς το πρώτο σκέλος των επιπλέον δαπανών. Ερώτηση δεύτερη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Φέρμ για τη θέση που έλαβε ως προς την άρση ε, των επιφυλάξεων και την απελευθέρωση του αποθεματικού. Και για τις ερωτήσεις σχετικά με τις μελέτες, χάρηκα τον κύριο Φέρμ να λέγει ότι ήταν ικανοποιημένος. Εγώ είμαι λιγότερο ε, ευχαριστημένος ακούγοντας την κυρία Γκρέσλε που είπε ότι δεν ικανοποιήθηκε πλήρως. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά πρόκειται για ε, ε, διοικητική αρχαιολογία για να σας δώσουμε τις ε, πληροφορίες που μας ζητήσατε. Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Πάρα πολύ σκληρή, επαναλαμβάνω, και σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα και να σας έχουμε στη διάθεσή σας όλες τις προφορίες που ζητάτε και σε πάρα πολύ μικρές προθεσμίες. Και μετά από τα διοικητικά θέματα που συζητήσαμε, θα κάνουμε όλοι προσπάθειες για να παραμείνουμε στο ιστορικό του τίτλου 5, έχοντας στο μυαλό μας και τις μεταφορές πιστώσεων. για να ανταποκριθούμε και στη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης. Λοιπόν, είναι Απόλυτος απαραίτητο να έχουμε στα χέρια μας όλες τις διαθέσιμες διοικητικές δαπάνες ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απευθύνω έκκληση, Πρόεδρε, στην Επιτροπή σας, τα κονδύλια αυτά να απελευθερωθούν δεδομένων των πλήρων ε, πληροφοριών που σας δώσαμε. Οι συνεργάτες μου λένε δεν ξέρουμε τι άλλο θέλετε, τι άλλο να δώσουμε άμα ζητήσουν κάτι επιπλέον. Σας έχουμε ενημερώσει εξαντλητικά. Αυτά ήταν τα δύο σχόλια και οι που ήθελα να θέσω υπόψη τη Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Merci beaucoup. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η Ζητώ συγγνώμη, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω το εξή στον κύριο Γενικό Διευθυντή. Στους ε, όρους και τις προϋποθέσεις για το αποθεματικό ήταν ήδη επικεφαλίδα και ο τίτλος της μελέτης. Δεν είναι έκπληξη Είναι εύκολο με τα προηγουμένα συστήματα πληροφορική ο υπάλληλο που το είχε αναλάβει να το δει. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ήταν προπόθεση και όρο. Δεν είναι καινούριο. Δεν βάζουμε νέα κριτήρια. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αφού το είχαμε ζητήσει ήδη από πριν. Ε, και έχει και λόγους αυτό που το ζητάμε. Πού πηγαίνουν τα κονδύλια αυτά για τις μελέτες, ποιες μελέτες, είναι σημαντικό ερώτημα και στα κράτη-μέλη μα τα ρωτάμε πάντα αυτά τα θέματα Στι κυβερνήσει Είναι 300 εκατομμύρια ευρώ αυτά που δαπανίσαμε για δαπάνε και νομίζω ότι έχει νόημα να μάθουμε ποιο πήρε τι και για ποιο λόγο. Και θα ήταν έτσι όμορφο και κομψό να μα τα δώσει αυτά τα στοιχεία. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ γκε. Ο Λάσλο. Λάσλο. Για συμπεράσματα. Παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε, πρέπει να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Σαλβαδόρ και Γιάννησεν για την υποστήριξή τους. Και ευχαριστώ τον Γκέρεν για τις παρατηρήσεις του. Σημειώνω διαφορά στάσεως μεταξύ ΕΛΚ και Σοσιαλιστών ως προς τις δημοσιονομικές υπηρεσίες. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συγγνώμη. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στις προτάσεις μας έχοντα συζητήσει και σύντομα με τον Σαλβαδόρ. Θεωρητικά θα ήθελα να πω ότι δεν μου αρέσει η ιδέα τα λεφτά αυτά να τα βάλω στην άκρη μόνο για έναν πελάτη. Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η πρόταση, θα ήταν διατεθειμένος ο εισηγητή σα να ε, κατανείμει ισομερός, ισοδίκαια τα ποσά αυτά, το ποσό αυτό στις 7 ε, όμοιες γραμμές του προπολογισμού. Πλην όμως τα χρήματα αυτά για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρέπει να πω ότι και περιορισμένα είναι και ως εκ τούτου εμείς έχουμε κατανέμει κατά αναλογία τα 10 εκατομμύρια τα 10 εκατομμύρια πάνω από το προσχέδιο και η αναλογία για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, θα έπεφτε στα 140 μόνο. Η αναλογία αυτή τώρα θα πρέπει να αλλάξει με βάση την πρόταση του Γκέραν για να φτάσει στις 700.000, δηλαδή 560.000 επιπλέον. Όπως είπα και από την αρχή, ως εισηγητής ε, εξετάζω το ενδεχόμενο να δεχθώ και την πρόταση της ολιστικής και της φιλελεύθερης ομάδας ε, και προτείνω να γίνει δεκτή αυτή η ιδέα. Οπότε και το περιθώριο, εάν μπορούμε να το πούμε περιθώριο αποθεματικό, θα είναι 146,747 ευρώ. Ευρώ, όχι εκατομμύρια, ούτε χιλιάδες. Μόνο ευρώ. Μηδέν δηλαδή. Πολιτικό μηδέν το αποθεματικό το περιθώριο. Όποιο δηλαδή θα κληθεί να μιλήσει στον τύπο, στο κοινό κτλ. Μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι μηδενικό το αποθεματικό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και ω εκ τούτου, γιατί να μην το κατανείμουμε στι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε σε κάποια άλλη γραμμή. Όπω είπα και νωρίτερα, καλύτερα να, να μην τα είχαμε κάνει τα χρήματα αυτά. Για σκεφτείτε τι θα συμβεί εάν μας λείψουν μερικές εκατοντάδες μετά από τον δεύτερο, τρίτο και τέταρτο έλεγχο. Για να το αποφύγουμε αυτό ενδεχόμενο λοιπόν και έχοντα πλήρη εμπιστοσύνη στη δουλειά τη Γραμματεία, σημειώνω ότι είναι ε, λογική αυτή η διασφαλιστική δικλίδα. Και η πρότασή μου είναι να διατεθούν επιπλέον 700 λέει ο μιλητή τη πρωτοπιστική Υπηρεσία. Μαζί με τα 140 που έχουν προγραμματιστεί και το επιπλέον 560. Και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει έτσι η γραμματεία. Και εκονάκων, ή εν πάση περιπτώσει, όχι με εκστασιασμένη χαρά. Ε, πιστεύω ότι θα μπορέσω να ακολουθήσω, θα μπορέσω να συμφωνήσω και πιστεύω ότι θα ακολουθήσει και το ΕΛΚΑ. Εν προκειμένου νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πω τα χρήματα ίσω είναι ψίχουλα, αλλά έχει μεγάλη σημασία η συνένεση και η αλληλεγγύη, η διάθεση να στηρίξουμε ένα τον άλλον. Αν και αυτό, όπω είπα από την αρχή, δεν είναι ιδιώδη λύση για μένα. Εν πάση περιπτώσει, για το μέσο μικροχρηματοδότηση. Ε, διάβασα εν συντομία τη σημειώσει από το τελευταίο διάλογο. Δεν είναι το πρόβλημα πραγματικό, αλλά αν αντιλαμβάνουμε σωστά την κατάσταση, υπήρχε συμφωνία ως προς τη δική μας πρόταση για το 2010. Και παραμένει λίγο πολύ εκρεμές ε, το μέλλον, η μοίρα της, ε, του μέσου μικροχρηματοδότησης. Ίσως θα μπορούσε η Επιτροπή να χρηματοδοτήσει εν μέρη από, το, από την πρόοδο και εν μέρη από φρέσκο χρήμα. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα εν προκειμένου, αλλά θέλω να πω το εξή. Ότι είναι λογικό να είναι δυνατόν μέσω μια νομική βάση να αποφασίζουμε για τα, για τα δημοσιονομικά θέματα, αλλά δεν είμαι βέβαιο εάν αυτό αποτελεί πάγια πρακτική, αν αποτελεί παράδοση και αν είναι και σόφρον λύση. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο να μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να διαφυλάξει αυτή την κατάσταση, αλλά δεν υπάρχει νομική βάση η οποία να επιτρέπει άμεση επέμβαση αριθμητική στους μελλοντικού προϋπολογισμούς. Άρα ό,τι και να αποφασίσουν εκεί είναι μόνο προσανατολισμός, τίποτε περισσότερο. Στο μέλλον, η Επιτροπή των Προπολογισμών και το Κοινοβούλιο στο σύνολό θα προσπαθήσουν βέβαια να ακολουθήσουν αυτέ τι τάσει, αλλά ποιο ξέρει με τι συνθήκε θα κληθούμε αργότερα να λάβουμε αποφάσει. Για δε την επικοινωνιακή πολιτική. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να καταπνίξω οποιαδήποτε πρόοδο και εργασία είχε γίνει σε επίπεδο της Γενικής Διεύθυνσης. Ε, είχα σαν στόχο να δώσω μηνύματα ότι βελτιώνουμε, ότι ενισχύουμε την επικοινωνιακή πολιτική και με τη Γενική Διεύθυνση την αλόγω γενική διεύθυνση, σε όλε μου τι συζητήσει, προσπαθώ να δείξω αυτό, ότι θέλουμε κάθε τι που θα κάνουμε να βελτιώνει την επικοινωνία μας, την επικοινωνική μας πολιτική. Εδώ λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε δεν είναι δημοσιονομικό και αν ε, μας πούνε ότι είναι ικανοποιητική η πρόοδος και τα στοιχεία που αναφέρονται στον προπολογισμό, δεν έχω παρά να δώσω το πράσινο φως. Επίσης για το τίτλο 5 αναφέραν ε, και ο συνάδελφος και άλλοι. Ε, πράγμα το οποίο είναι παράδοξο, γιατί δεν ήταν καθόλου εύκολο στη συνδιαλλαγή να δεχθούμε την ιδέα ότι η Επιτροπή μπορεί να γνωρίζει ότι χρειάζονται περίπου 80 εκατομμυρία για την ε, αναπροσαρμογή των μισθών, αλλά και ότι το γνωρίζει δεν τα ζητεί αυτά τα 80 εκατομμύρια, γιατί είναι πεπισμένη ότι κάθε θεσμικό όργανο έχει ένα κρυφό αποθεματικό όπως θα το λέγαμε. Εμείς δεν είμαστε πεπισμένοι όμω ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Και ω εκ τούτου, η λύση, η φόρμουλα που έχουμε βρει για τον ε, τίτλο υπαριθμών 5 είναι να λάβουμε υπόψη αυτή την εξέλιξη και να προστατεύσουμε, να δεν φυλάξουμε το παθηματικό για τη Λισαβόνα, όπως αναφέρεται μέσα στον τίτλο. Αν και δεν ήμασταν ε, σε θέση να βρούμε αυτά τα επιπλέον 80 εκατομμύρια τώρα. Ή εν πάση περιπτώσει δεν πιστεύουμε την Επιτροπή. Σας είπα ότι είναι παράδοξη η κατάσταση. Δεν ξέρω πώ Σα να είναι δυνατόν κάτι τέτοιο, δεν μπορώ να το φανταστώ, αλλά φαίνεται ότι είναι πεπισμένη η Επιτροπή ότι είναι δυνατόν να διαχειριστεί την κατάσταση κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα αποδεικνύεται όμω ότι είναι υποχρεωτική η αναπροσαρμογή των μισθών. Ε, δεν ξέρω κύριο Σέλης, αν θα συμφωνήσει ότι το ποσοστό είναι 3,7% για την αύξηση. Ασχέτως των προθέσεων των ΜΕΝ και των ΔΕ υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν διατάξεις. Και αν έχω καταλάβει καλά την υπόθεση, υπάρχουν δύο δεδομένα. Αφενός μεν το ποσοστό του πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει ο μιλητής, στις Βρυξέλλες, δεν ξέρω με ποιο όρο, με, με ποιο γεωγραφικό χώρο οριοθετείται και ταυτόχρονα η εξέλιξη των μισθών στις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, που επίσης έχουν κάποια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Άρα τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να επικρίνουν εμάς, γιατί μπορεί τώρα να παγώνουν τα κράτη-μέλη, αλλά αυτό θα έχει επίπτωση στους μισθού στην αναπροσαρμογή του χρόνου. Όλα αυτά όμω να λύσουν Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν από ό,τι βλέπω να ε, εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Ε, τώρα όμως δεν υπολογίζεται ένα, ούτε ένα ευρώ ως ε, προσαρμογή, αναπροσαρμογή με το 2010. Από ό,τι φαίνεται θα το διαχειριστεί το θέμα αυτό το κάθε θεσμικό όργανο χωριστά. Εν τέλει, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του άλλου συναδέλφου που μίλησαν για την υποστήριξη που μου προσέφεραν και θα ήθελα να μάθω ή μάλλον να σας πω ότι στο συμπληρωματικό φάκελο υπάρχει η περιληπτική ανάπτυξη του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Τα στοιχεία όμως ε, όσο και αν δεν είναι πολύ ενδιαφέροντα, γιατί έχουμε τις σταθερές τιμές του 2004 που έχουν μεταξύ εξελιχθεί. Όμως τα ποσοστά του ακαθάριου εγχωρίου προϊόντος είναι, εθνικού προϊόντος είναι ε, ενδιαφέροντα, είναι σαφή και έχουμε συνολικές δεσμεύσεις υποχρεώσεων 1,06. Εμείς είχαμε συμφωνήσει 1,2. Το ξεπερνάμε λοιπόν. Επίσης η εκτίμηση πρόβλεπε καταβολή ε, μια ποσοστιαίας μονάδας. Εμείς δώσαμε 1,4. Άρα μπορούμε νομίζω να έχουμε έναν λογικό αλλά και σχετικά ε, πλούσιο προϋπολογισμό, μεγάλο προϋπολογισμό δεδομένων και των ε, περιόδων των εποχών που ζούμε. Και πρέπει, Πρόεδρε, να πω ότι το μήνυμα εξ αρχή ήταν ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι μέρος του προβλήματος. Μπορεί να αποτελεί έναν από τους λόγους της κρίσης, ε, μάλλον τα αποτελέσματα της κρίσης, αλλά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για να αποτελέσει μέσω επίλυσης ή αντιμετώπισης της κρίσης, εάν αξιοποιήσουμε σωστά τα χρήματα αυτά. Αυτό είναι ένα στόχο τον οποίο θα πρέπει να επιδιώξουμε μακροπρόθεσμα και όλα θα πρέπει και οι συνάδελφοι να επιδιώξουμε καλύτερη ενημέρωση, καλύτερη γνώση, ταχύτητα, στόχευση, αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα της δήλωση αυτής είναι ότι καλούμε τα κράτη-μέλη να επαναξιολογήσουν τα τρέχοντα προγράμματα ε, αξιολόγησης και να αξιοποιήσουν τα χρήματα και για την ανοίξη του ΑΕΠ και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την ανάπτυξη δηλαδή και όχι για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να περιμένουν και να γίνουν αργότερα. Ε, όπω σε παραδείγματα ανοικοδόμηση πόλεων και τα λοιπά Πράγματα που είναι πολύ ωραία μένα, αλλά δεν επήγουν τώρα. Η πραγματική οικονομία χρειάζεται υποστήριξη και αυτό είναι ο στόχο τη δήλωση. Αυτό το στόχο εξυπηρετεί η δήλωση και ελπίζω να την υποστηρίξουμε όλοι. Ελπίζω να προσδορίσουμε στο τέλος ε, την ώρα τη ψηφοφορία την ε, στάση μας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες, όλα τα κείμενα on block. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Νομίζω ότι σε λίγα λεπτά πολύ γρήγορα μπορούμε να τα ολοκληρώσουμε και να τα αποφασίσουμε αυτά στους συντονιστές. Η πρότασή σας για τη χρηματοδότηση, η τροπολογία δηλαδή για τα νέα ε, χρηματοπιστωτικά όργανα, οδήγησε σε συνένεση από πλευρά του συντονιστού των σοσιαλιστών που ε, ένευσε θετικά. Το ΕΛΚ λίγο, πώς να το πω, έκανε μια γκριμάτσα σαν να του είχαν δώσει μουρονόλαδο με το ζόρι να το φάει. Αλλά ξέρουμε ότι το μουρονόλαδο κάνει καλό στην υγεία όσο δυσάριστο και να είναι στη γεύση. Ε, θα ε, συμφωνήσουμε, είμαι βέβαιος. Λοιπόν, σας προτείνω να ολοκληρώσουμε εδώ αυτή την ανταλλαγή απόψεων για τα διάφορα στοιχεία της δεύτερης ανάγνωσης, δίνοντας το λόγο στο Ράιμερ Μπέγκε, που είναι ειδικό συζητητής για το δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο ευελιξίας και τα δύο δηλαδή αυτά τα θέματα για την ενδιάμεση θεωρήση και την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας. Και για τα δύο αυτά ο Ράιμερ έχει ε, συντάξει ένα έγγραφο εργασίας και επειδή η συμφωνία στη συνδιαλλαγή για τη χρηματοδότηση του προπολογισμού του 2010 συμπεριλαμβάνει τροποποίηση των δημοσιονομικών προοπτικών, καλά θα κάναμε να δούμε πιο μακροπρόθεσμα πώς εγγράφεται η συμφωνία αυτή στο συνολικότερο πλαίσιο. Λοιπόν, Ράιμερ, αν θέλεις να μας παρουσιάσει και τα δύο στοιχεία μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά αυτό που μου ζητάτε, πρέπει να μιλήσω και για τις δύο εκθέσεις. Κινητοποίηση του μέσου βελεξίας και τα μελλοντικά, έτσι, για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Όντως, οι δύο πρώτες ε, εκθέσεις έχουν ε, σχέση με το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής του προπολογισμού. Το μόνο που θα ήθελα να σας πω είναι ότι στο ψήφισμα ή στα ψηφίσματα έχω επαναλάβει ότι για το μέσο ευελιξίας καταφέραμε να επιβάλλουμε 195 εκατομμύρια επιπλέον στα πλαίσια της δημοσιονομικής αυτής περίοδου, πρέπει να σας πω, της προγραμματικής, τρεις αναθεωρήσεις είχαμε και για την ευελιξία ε, και το συνολικό ποσό μαζί με το Γαλιλαίο και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, ε, την επίγουσα βοήθεια και την ε, ανάκαμψη έχουμε φτάσει στα 8,4 δισεκατομμύρια στο μεταξύ. Ε, σε τρεις διαδικασίες για τον προπολογισμό χρειάστηκε να τα επιβάλλουμε, να τα προσθέσουμε ε, με τα μέσα που μας δίνει η διοργανική ε, συμφωνία. Στο ψήφισμα 6 έχω κείμενο συγγνώμη, του ψηφίσματος έχω πει ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια. Η χρηματοδότηση της ασφάλειας ε, του Κοσλοντούι δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε θυσίες στα προβλήματα προγράμματα της κατηγορίας 1α. Δεν είναι αυτόματο δηλαδή ότι θα πρέπει να πληγούν αυτοί. Υπάρχουν και άλλα θέματα προς συζήτηση και στο ψήφισμα για την αλλαγή του δημοσιονομικού προγραμματισμού στο σημείο 6 αναφέρω στα αγγλικά θεωρεί ότι το παρόν πλαίσιο δεν μπορεί να καλύψει όλε τι ανάγκε χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό καλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πρόταση για την ενδιάμεση αναθεώρηση ε, για το τρέχον πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο το συντομότερο. Αυτό θα το δούμε και αύριο στη συζήτηση και στη ψηφοφορία της έκθεσης ε, Σόριαν. Ε, αν κατάλαβα καλά από τροπολογίε, τροπολογίες, αυτό έχει συμπεριφθεί. Ο Τζέιμ Έλλη ρώτησε προηγουμένω τι γίνεται τώρα με την ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου και τι ζητάω εγώ και πώς μπορεί κανείς να προετοιμαστεί. Αναφέρεται μάλλον στο 3.6 στην τελευταία παράγραφο του δικού μου κειμένου για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Τώρα όμως δεν ξέρω ποια είναι η δική του διαδικασία. Διαβάζει όλο το κείμενο ή αυτό που έκανα παλαιότερα εγώ στα αστυνομικά διάβαζα πρώτα το τέλος και μετά ξανά από την αρχή. Βέβαια, όταν μιλάει κανείς για πολιτικές προτεραιότητες και προσανατολισμό μιας νέας επιτροπής και το, όταν το συζητάει με τον υποψήφιο, ακόμα και αν το γνωρίζουμε σχετικά καλά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ακρόαση για να δούμε και τα παράλληλα θέματα που συζητούμε για διοργανικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κέντρα βάρους και όλα αυτά που κάποια στιγμή ε, θα αποφασίσουμε από κοινού να κάνουμε συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ε, και ε, επιτρέψτε μου να πω σε 30 δεύτερα ότι θα πρέπει μόνοι μας να ασχοληθούμε με αυτό το έργο και ε, όχι όπως έγινε σε άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή με κάποια μελέτη, δεν ξέρω, αναθέσανε σε think tanks, σε ομίλους προβληματισμού για να δούμε τι έγινε στην Επιτροπή τα τελευταία πέντε χρόνια, ποιες ήταν οι πολιτικές προτεραιότητες για το επόμενο διάστημα και σε ένα τρίτο κεφάλαιο, πάλι με think tank, δίνουν τις ερωτήσεις να κάνουν στους επιτρόπους. Ποιες είναι οι σωστές ερωτήσεις για τους υποψηφίους επιτρόπους για να δώσουν και τις σωστές κατευθυνόμενες απαντήσεις. Από ό,τι φαίνεται αυτό έκανε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, παρακαλώ. Ε, να τα χρήματα για τις μελέτες. Καλύτερα θα πήγαιναν αλλού και θα πιαναν τόπο περισσότερο. Αλλά είναι αυτοτελείς και αυτόνομες οι επιτροπές και εγώ αγωνίστηκα πάντα ε, γι' αυτό να αποφασίζουν κυρίαρχα πού θα δίνουν τα χρήματα. Αυτά εισαγωγικά τώρα. Βεβαίως έχουμε και μια σύγχυση ως προς τους ορισμούς. Τι θα πει ενδιάμεση να θεώρησε ο καθένας, καταλαβαίνει ίσως κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει νόημα να θυμίσουμε αυτό που είχε γίνει όταν αποφασίστηκαν ε, οι δημοσιονομικές προοπτικές και τι ε, δηλώσεις είχαμε κάνει τότε και τι είπε το κάθε θεσμικό όργανο. Και τι εννοεί δηλαδή το κάθε θεσμικό όργανο με όλα αυτά. είχε υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είχε αναλάβει την υποχρέωση, δηλαδή να καταθέσει έκθεση περί τα τέλη του έτους 2009, αυτό το καιρό δηλαδή, και αν χρειάζεται και να καταθέσει αντίστοιχε προτάσεις. Από εκεί και πέρα, με βάση τα όσα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2005 για τα συμπεράσματα, ε, καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ευρύτατη αναθεώρηση, review ή revision ανάλογα με το κείμενο, αναφέρεται διαφορετικά, για την πολιτική δαπανών μεταξύ αυτών και τις γεωργικές δαπάνες και τη Βρετανική επιστροφή. Για όλα αυτά το 2008-2009. Και αυτή η αναθεώρηση, αυτό το συμπληρώσαμε εμείς, θα πρέπει να ε, έχει και μια αξιολόγηση για το πώς λειτουργεί η διοργανική συμφωνία. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση ίσως, γιατί ε, το 2008-2009 ε, να γίνει αξιολόγηση και να συνδέσουμε τις γεωργικές δαπάνες, τη Βρετανική επιστροφή με τη διοργανική συμφωνία και το 2009 ε, είναι λίγο πίεση χρονικά αυτό γιατί ξέραμε ότι θα τεθεί ε, αργότερα σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας για λόγους γνωστούς σε όλους μας και καταλάβαμε ότι όλα αυτά θα συμπέσουν χρονικά. Λοιπόν, ε, είχαμε δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας τότε στο Κοινοβούλιο, μία για την ενδιάμεση αναθεώρηση το Μάρτιο, την οποία έκθεση κατέθεσα εγώ τότε, σε στενή πάντα συνεργασία και συνεννόηση με την Κατρίν Γκικέν για ε, τις ε, δημοσιονομικές ψυχές της συνθήκης της Αβώνας που ακολούθησε στην Ολομέλεια αλλά είναι πολύ στενά συνδεδεμένες οι δύο εκθέσεις και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τις δημοσιονομικές τους συνέπειες. Είναι βεβαίως σαφέστατο ότι τότε συνδέθηκε πολύ και ε, το θέμα της διοργανικής συμφωνίας και το τι σημαίνει ε, για τα εργαλεία και τα μέσα που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους πλέον τα θεσμικά όργανα μετά τη Λισαβόνα για να ασκούν μια επιτυχή δημοσιονομική πολιτικής. 25 Μαρτίου 2009 ενέκρινε η Ολομέλεια την έκθεση αυτή και βάσει του εγγράφου εργασίας που λέγει ότι θέλουμε μια σταδιακή προσέγγιση σε τρία στάδια δηλαδή. Πρώτον, να δούμε, να εντοπίσουμε ποια είναι τα ελλείμματα και τα πολυφάδια ε, της ε, δημοσιονομικής προοπτικής και, και στα πλαίσια του ενεάυσιου χαρακτήρα του προεπολογισμού και ε, αν γίνεται να αλλάξει αυτό με μεγαλύτερη ευελιξία και αν είναι αναγκαίο με χρήση των ε, αποθεμάτων κάτω του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων. Αυτή ήταν η τότε ε, διατύπωση. Επίσης, και ταυτόχρονα είπαμε ότι έχουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση των διαφόρων πολιετών προγραμμάτων και μπορούμε να την αξιοποιούμε. Έχουμε 50 με 60 πολυετή προγράμματα στη συναπόφαση σε μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία και το 2010 και το αργότερο το 2011 τα περισσότερα προγράμματα αυτά βρίσκονται στο ίμιση της ε, ζωής τους και θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση ενδιάμεση τι λειτουργεί καλά, τι λειτουργεί λιγότερο καλά, που χρειάζονται προσαρμογές, που χρειάζονται αλλαγές γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε χρόνια ολόκληρα μέχρι ε, ότου να συζητήσουμε αυτές τις αλλαγές για να τις επιβάλλουμε. Χρειάζεται λοιπόν και κάποια συνέχεια αφενός, αλλά αφετέρου ε, εγκαίρως να θέσουμε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων όταν αυτό χρειάζεται. Άλλο θέμα που είχαμε πει τότε. Ήταν και τμήμα άλλωστε αυτού του πολιτικού συμβιβασμού. Λέμε λοιπόν, αν ε, γίνεται λόγος πλέον για ενδιάμεση αναθεώρηση και γνωρίζουμε ταυτόχρονα ότι κατά πλειοψηφία τότε τουλάχιστον και η Επιτροπή και το Συμβούλιο όταν μιλούν για αναθεώρηση, review δεν εννοούν τίποτα διαφορετικό παρά προετοιμασία των επομένων δημοσιονομικών προοπτικών από το 2014 και μετά. Ε, τότε γνωρίζουμε ότι αυτή η άσκηση είναι πάρα πολύ δύσκολη ενδιάμεση αναθεώρηση για την τωρινή προγραμματική περίοδο που είναι 2007 με 2013 και ταυτόχρονα σχεδόν αρχίζουμε να συζητάμε και να προγραμματίζουμε ε, τα πρώιμα στάδια της ε, προγραμματικής περίοδου μετά το 2014. Και σε στενή πάντα συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καταλήξαμε στο να πούμε ότι ας κάνουμε μια προσφορά Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ελλείμματα. Γνωρίζουμε ότι χρειάζονται προσαρμογή τα μέσα και τα όργανα που έχουμε στη διάθεσή μας για να δρούμε πιο γρήγορα και πιο ευέλικτα και να μην ε, χρειαστεί αυτός ο στραγγαλισμός για να φτάσουμε στα 8,4 δις. Και έχουμε και τη συνθήκη της αγώνας που έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις και αυτό όλα θα πρέπει να ενταχθούν στην πολιετή δημοσιονομική πολιτική μας. Ωραία. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι πολλά μέλη στο Συμβούλιο αποφεύγουν όπως ο διάβολος στο λιβάνι αυτές τις διαδικασίες αναθεωρήσεις, αναπροσαρμογές και ανακατατάξεις. Γι' αυτό είπαμε τότε. Ωραία, τότε να παραμείνουμε στην αναθεώρηση, φιλόδοξη όμως, Λισαβόνα και τα συμπαραμαρτούντα, για παράδειγμα ένα ταμείο για την προστασία του περιβάλλοντος και κατά της κλιματικής αλλαγής και αυτό ε, είναι και στην επικαιρότητα και το έχουμε σκεφτεί. Ήδη από το Μάρτιο το βλέπαμε και το έχουμε στο ψήφισμά μας. Λοιπόν, και να το συνδέσουμε μετά με την προσφορά ότι αν πετύχουν όλα αυτά και πείσουμε ε, το Συμβούλιο και την Επιτροπή δια της πυθούς αλλά και δια του πείσματος να επιτύχουμε ε, παράταση μέχρι το 2015 2016 του παρόντος συστήματος και της προγραμματικής περίοδου. Και μετά να αρχίσει το επόμενο στάδιο με τη νέα δημοσιονομική περίοδο, προγραμματική περίοδο που να αρχίζει το 2016-2017 και να συνδέεται και με την εντολή και τη θητεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και η Συνταγματική Επιτροπή το ψήφισε. Τότε την έκθεση την είχε ο συνάδελφος Δεχάνε. Γιατί είναι ένα δημοκρατικό έλλειμμα αυτό. Πάντα έχουμε το Κοινοβούλιο που πρέπει να διαπραγματεύεται για ένα πολιετές ε, πρόγραμμα. Τελικά τις συνέπειες ε, ε, τις λούζεται το επόμενο Κοινοβούλιο που δεν ήταν σε θέση να διαπραγματευτεί τα όσα το δεσμεύουν, το διέπουν και είναι περίπου το, το, ελισοδεμένο το κοινοβούλιο το επόμενο πάντα, χωρίς να είχε την ευκαιρία να διαπραγματεύεται όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για τις επιμέρους κατηγορίες του προπολογισμού και τους τίτλους και τους κλάδους και τους τομείς, για τις νομοθετικές βάσεις, για τις νομοθετικές βάσεις, ή για κάποιες προθεσμίες και διάρκειες ε, διαφόρων κατηγοριών και τίτλων του προϋπολογισμού. Δηλαδή δεν είναι σημειολογική τώρα αυτή η συζήτηση, τι είναι mid-term review και review of the budget, ενδιάμεση αναθεώρηση δηλαδή και ε, η αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Μπορεί χρονικά να έχουμε κάτι διαφορετικό στο μυαλό μας από αυτό που εννοούσαμε μέχρι τώρα ή εννοούσε το Συμβούλιο και η Επιτροπή και συζητούσε στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Και εδώ θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ήδη από την αρχή του επομένου έτους να δούμε ποια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ε, ζητάει τι θα κάνουμε εμείς στην έκθεσή μας, τι θα κάνουμε την πρόταση για τη δημιουργία της εξωτερικής ε, δράση τη Υπηρεσία. Τι κάνουμε με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου ο πολιετής προγραμματισμός θα πρέπει να περάσει τώρα σε ένα πολιετές ε, χρηματοδοτικό πλαίσιο υπομορφή νόμου και συμφωνία του Κοινοβουλίου πριν αποφασίσει το Συμβούλιο. Αυτή η προσαρμογή προβλέπεται στο άρθρο 304 της Διοργανικής Συμφωνίας. Έχουμε εδώ την συναπόφαση, έτσι. Αλλάζει η κατάσταση και ποιοτικά αλλάζει για το Κοινοβούλιο. Και επίσης έχουμε κάποια στοιχεία της ε, της Ρωμανικής συμφωνίας που είναι απαρχιωμένα και θα καταργηθούν. Υπάρχουν άλλα στοιχεία που παραμένουν και κάποια άλλα που λόγω των νέων δομών χρειάζονται νέα διαπραγμάτευση ε, ή συμπλήρωση, εν πάση περιπτώσει. Διότι ε, οι πολιτικές συνθήκες ε, το επιβάλλουν ε, λόγω της συνθήκης της Αβώνας. Να δούμε πώς θα ε, γίνει αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης, η διπλωματική υπηρεσία. Πώς θα διαρθρωθεί αυτό το σώμα, γιατί ανάλογα με αυτό υπάρχουν προγράμματα εξωτερικής δράσης που χρειάζονται αναπροσαρμογή ή μεταφορά πιστώσεων ακόμα όταν έχουμε και μεταφορά αρμοδιοτήτων από το την Επιτροπή στην ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι μεγάλο το πακέτο αυτό, όντως πολύ φιλόδοξο και γι' αυτό δεν θα πρέπει να κάνουμε την ε, κίνηση, το σφάλμα μάλλον, να ε, διαπραγματευτούμε κάτι χωρίς να έχει καταλήξει κάτι άλλο. Γιατί θα αποδυναμωθούμε, δηλαδή να μην περάσουμε στο δεύτερο στάδιο των διαπραγματεύσεων πριν ε, ξεκαθαρίσει το πρώτο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι από την άποψή μου, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πολιτικά, θα πρέπει να πάμε στις διαπραγματεύσεις με μία προσέγγιση που να μην ε, μας ικανοποιεί η μινιμαλιστική λογική. Παρόλο που γνωρίζουμε ότι τώρα δεν είναι εύκολο αυτό για τα κράτη-μέλη, και δεν σας κρύβω ότι τις τελευταίες μέρες διάβασα και μελέτησα την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και πρέπει να σας πω ότι είναι αυτονόητο ότι έχω προβλήματα ε, να ζητήσω περισσότερα χρήματα όπου το φανάρι του ελεγκτικού συνεδρίου είναι στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο. Θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται και ε, να φροντίσουμε να απλοποιούμε τις διαδικασίες γιατί βλέπουμε στο ελεκτικό συνέδριο να ανάβουν κόκκινα λαμπάκια και να χτυπάνε καμπανάκια. Θα πρέπει να τα λύσουμε αυτά πριν συζητήσουμε για νέα χρηματοδότηση. Αυτή λοιπόν η ενδιάμεση αναθεώρηση τελικά θα πρέπει να καταδείξει ότι το Κοινοβούλιο προσπαθεί να παίξει το ρόλο του συνειδητά ως ε, δημοσιονομική αρχή με τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά επίσης θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι προφανώς δεν θα πρέπει από τη μια μέρα στην άλλη, δεν μπορούν από τη μια μέρα στην άλλη να τεθούν σε ισχύ όλες οι χρηματοοικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της Λισαβόνας και εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια σταδιακή μετάβαση. Βλέπε διάστημα, βλέπε ενεργειακή πολιτική πέρα από τη διπλωματική υπηρεσία, βλέπε συνεργασία στη δικαιοσύνη. Όλα αυτά σημαίνουν και κονδύλια του προϋπολογισμού για να υλοποιούνται. Για να είμαστε τελείως γυμνοί ε, σε αυτούς τους τομείς πολιτικής. Και το παλιό κοινοβούλιο είχε ήδη αποφασίσει αυτή τη σταδιακή ε, πορεία Να μην απογειωθούμε δηλαδή, να αφήσουμε σιγά σιγά ε, να ε, παρασυρθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και να τα έχουμε υπόψη μας όταν μιλούμε για τις συνέπειες της συνθήκης της Σαββόνας και πώς υλοποιούνται στην πράξη αυτά και πώς μεταφράζονται σε οικονομικούς όρους για να μπορέσουμε και σε αυτή τη συζήτηση θεσμικά να είμαστε στο πλευρό του Κοινοβουλίου και όχι στο πλευρό του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Bien, merci, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής και εξαντλητική η παρουσία σου και επομένως ε, ήσουν πάρα πολύ σαφής και νομίζω ότι θα ξέρουμε και τι να ρωτήσουμε στην ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα και από πολιτική και από πρακτική άποψη και να τα διαχειριστούμε πρακτικά έτσι ώστε να εκπονήσουμε το κατάλληλο χρονοδιάγραμμα. Είμαστε όλοι βετεράνοι εδώ βέβαια για τα ευρωπαϊκά θέματα και ξέρουμε ότι όταν συμφωνούμε για την ε, ημερήσια διάταξη και για το χρονοδιάγραμμα έχουμε κάνει την περισσότερη δουλειά. Επομένως, η διαπραγμάτευση θα αφορά πρώτα το χρονοδιάγραμμα και βεβαίως το περιεχόμενο, δηλαδή ποια είναι τα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε και ποιες είναι οι νέες ανάγκες που θα λάβουμε υπόψη μας. Και φυσικά δουλεύουμε μετά πάνω σε προτάσεις της Επιτροπής και είναι ακριβώς η ανταλλαγή απόψεων που θα πρέπει να έχουμε με τον υποψήφιο Επίτροπο. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και πολλές αποφάσεις οι οποίες αποτελούν μία ενιαία δέσμη η οποία θα πρέπει να συμφωνηθεί πολιτικά επανειλημμένα μία, δύο, τρεις φορές που όμως ε, πρόκειται για αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στη διάρκεια του έτους 2010 όσον αφορά την θεσμοθέτηση των νέων θεσμών με νομική βάση, την υλοποίηση νέων πολιτικών ή την διεύρυνση αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις απαραίτητες νομικές βάσεις δηλαδή τι σημαίνει ε, ε, αρμοδιότητα όσον αφορά τα ενεργειακά, τι σημαίνει όσον αφορά το διάστημα κτλ. Ο Ράινερ μας έδωσε και κάποια παραδείγματα. Η πιστώσεις ε, που είναι απαραίτητες έτσι ώστε να δοθεί ένα περιεχόμενο σε αυτές τις αρμοδιότητες και έτσι ώστε να υπάρξει η νομική βάση. Βεβαίως, ε, θα χρειαστεί νέα τροποποίηση των δημοσιονομικών προοπτικών. Πρόκειται για αναθεώρηση, ε, πρόκειται για απλή προσαρμογή. Η Επιτροπή θα κάνει την πρότασή της. Αλλά με βάση ποια διαδικασία, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει συγκεκριμένο καθεστώς για τις πολιετής ε, ε, προβλέψεις που μέχρι τώρα είχαν ένα ιδιαίτερο περίεργο νομικό καθεστώς, ένα είδος συμφωνίας ε, που έπρεπε να ε, έχουν τα τρία θεσμικά όργανα. Ενώ τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο ε, καθεστώς, νομικό καθεστώς υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου. Και επομένως θα πρέπει να δούμε αν πρόκειται εδώ για μια τροποποίηση ή για την ε, ουσιαστική εφαρμογή του πραγματικού πολιετούς προγραμματισμού μετά το 2014. Στις ε, πρώτες επαφές ε, με την ε, Ισπανική Προεδρία κατάλαβα ότι θα ήταν ιδιαίτερος ευτυχής η Ισπανική Προεδρία εάν εάν δεν συζητούνται τα ζητήματα αυτά. Αλλά βεβαίως ε, εμείς δεν είμαστε εδώ για να δίνουμε χαρά και ευτυχία στην Ισπανική Προεδρία και από την άλλη πλευρά, μην ξεχνάμε ότι για τον προπολογισμό του 2011 θα ακολουθηθεί η διαδικασία της Λισαβόνας και επομένως ε, ε, σύμφωνα με τη διαδικασία της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Επίσης, πολύ σωστά το παρουσίασε ο Ράιμερ και διαπιστώνουμε λοιπόν, βάσει και της παρουσίασης αυτής, ότι το πρόγραμμα εργασίας και η επιλογή του χρονοδιαγράμματος ε, και των προτεραιοτήτων, των χρονικών προτεραιοτήτων είναι το σημείο εκκίνησης το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει από πολιτική άποψη. Είναι το, το σημείο πολιτικής εκκίνησης αν θέλετε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα η πολιτική εξόδου της, ε, από την κρίση. Μετά από τα προγράμματα ανάκαμψης, τα οποία καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε το 2010, θα χρειαστεί πολιτικά, κοινοτικά, νομικά εργαλεία και κυρίως θα απαιτήσει πολιτικά μέσα, δημοσιονομικά μέσα, νομικά μέσα σε εθνικό επίπεδο, όπως ακριβώς έγινε και τη στιγμή της αντιμετώπισης της κρίσης και βεβαίως εδώ παίζει ύψιστο ρόλο ο πρόεδρος, ο προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και πέρα από την νέα ΚΕΠΑ που θα προταθεί από τον ύπατο εκπρόσωπο ε, θα υπάρξουν και κάποιες νέες απαιτήσει. Και βεβαίω να πούμε, και ευχαριστήσουμε τον Ράιμερ για το έγγραφο που μα υπέβαλε, να πούμε ότι η Επιτροπή Προπολογισμών, η Επιτροπή μας πρέπει να έχει μια γενικότερη έποψη των θεμάτων που θα βρεθούν απέναντί της, των θεμάτων και των ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει όταν θα έρθει η στιγμή βεβαίως. Έχω δύο αγόρτες που έχουν ζητήσει τον λόγο, Έινερ και μετά ο Τζέιμς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο μόνο για να κάνω μια εκτίμηση, αξιολόγηση του εγγράφου εργασίας που μας παρουσίασε ο κύριος Μπέγκε για να δούμε πώς θα μπορούσε στο μέλλον να προσανατολιστεί η δουλειά μας. Βασικά συμφωνούμε με τις ιδέες του κειμένου. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι η σημασία της γλωσσικής απόχρωσης και της διαφοράς ανάμεσα στο ε, review και στο revision το εξήγησε ο κύριος Μπέγκε και το καταλαβαίνουμε και εμείς γιατί πολλές φορές κάναμε τροπολογίες για την έκθεση Σούριαν για τον προπολογισμό του 2010 της Ένωσης. Επίσης θα θέλαμε να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και λογικό κυρίως οι δημοσιονομικές προοπτικές να είναι πενταετούς διάρκειας και να μην είναι μόνο πενταετούς αλλά να συμπίπτουν χρονικά με ε, τη θητεία του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για ποιο λόγο. Δεν είναι δυνατόν εμείς να αποφασίσουμε για δημοσιονομικές προοπτικές που στη συνέχεια θα πρέπει να διαχειρίζεται το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι δημοσιονομικές προοπτικές επταετούς διάρκειας είναι κατά την άποψή μου υπερβολικά ε, μεγάλο διάστημα. Εμείς τώρα έχουμε δημοσιονομικές προοπτικές από το 2004, που είναι πολλά χρόνια πριν. Λοιπόν, να, μην είναι επταετής η διάρκεια. Και το 2004 τώρα θα πάει μέχρι το 2014, 10 χρόνια. Και ε, αυτές τις μέρες βλέπουμε ε, να δυσκολεύεται το Συμβούλιο και ακόμα και στην αναθεώρηση και δεν είναι καθόλου πρακτικά αυτά τα ζητήματα. Επίσης, Αυτό που μας απασχολεί σήμερα, η διάμεση αναθεώρηση, είναι κάτι που αποφασίστηκε στην προηγούμενη θητεία. Εμείς δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στο επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Καλό θα ήταν λοιπόν το παρόν Κοινοβούλιο να αποφασίσει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να την κάνει την αναθεώρηση και για ποιο λόγο. Από αυτή την ιδέα να ξεκινήσουμε. Και κάτι άλλο που με εκπλήσει, δεν ξέρω ε, ίσως θέει που είμαι καινούρια. Γιατί υπάρχει αυτή η επιφύλαξη, αυτός ο δισταγμός. Ενδιάμεση αναθεώρηση δεν σημαίνει εκβάθρον αναθεώρηση. Σημαίνει να κοιτάξουμε τι δεν πήγε καλά, να κάνουμε κάποιες προσαρμογές όπου χρειάζεται για να λειτουργήσουν καλύτερα ή να προσθέσουμε νέα τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τη θέση ισχύ της συνθήκης της Αβώνας και τις νέες προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Μου διαφεύγει πάρα πολύ γιατί υπάρχει αυτός ο δισταγμός, αυτό το κούμπομα για την ενδιάμεση αναθεώρηση. Και μια ερώτηση. Να δω αν θα μου απαντήσετε γιατί μου μπήκε μια αμφιβολία. Εμείς θα εγκρίνουμε το δημοσιονομικό κανονισμό και για πρώτη φορά θα βάλουμε εκεί το δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι, που είναι τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας. Ωραία. Αλλά τώρα έχουμε προοπτικές από το 2007 στο 2013. Δεν νομίζω ότι θα είχε νόημα σε έγγραφο του 2010 να μπει κάτι που αποφασίστηκε το 2007. Αλλά και πάλι δεν μπορούμε να πούμε περίοδος 2010 με 2013. Γιατί λέμε το ελάχιστο είναι πενταετής διάρκεια. Μήπω λοιπόν χρειάζονται αναθεώρηση δημοσιονομικές προοπτικές από το 2015-2016 να αφορά αυτό και το επόμενο κοινοβούλιο. Αυτά και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, James. Ευχαριστώ. Αλλά και πάλι έχω τρεις απλές ερωτήσεις. Πριν από τις εκφράσεις. Είναι δυνατόν, ίσως από τη γραμματεία των προπολογισμών, να ενημερωθούμε για το τι αλλαγέ θα επιφέρει η συνθήκη τη Λισαβόνα στον προπολογισμό, τις διαδικασίες, την ε, λογοδοσία προς τις ε, πολιτικές ε, στα εξωτερικών, των εξωτερικών σχέσεων. Γιατί ακούγονται διάφορα για το ότι θα πρόκειται μια συνεργασία μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου ή υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ποιος θα διαχειρίζεται τον το εκπρόσωπο, τη θέση του είπα του εκπροσώπου κτλ. Καλό λοιπόν θα είναι να είμαστε ξεκάθαροι, να ξεκάθαρη κατάσταση προ την υποχρέωση λογοδοσία πριν αρχίσουμε να δαπανούμε τα χρήματα. Επίση, είπατε νωρίτερα ότι κοτέ ερωτήσει λαμβάνουν κουτέ απαντήσει. Ξέρω πολύ καλά τι εννοείται, γιατί ποτέ δεν είναι σαφέ από πού προέρχονται αυτέ οι ερωτήσει ή τι, ε, σε τι μπορεί να αποσκοπούν. Όσο, όσο είναι σκόπιμο ίσω να διατυπώσουμε τι ερωτήσει αυτέ, γιατί ο κάθε ή, ε, ή κάθε επιτροπός θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των κονδυλίων που δαπανά και δημόσια μάλιστα να λογοδοτούν από την άλλη προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί Μπορεί να υπάρχει παρακολούθηση και το monitoring των προπολογισμών για αρκετά χρόνια, αλλά όταν είμαστε σε θέση να ζητήσουμε συγκεκριμένους λογαριασμού τότε μπορούμε να κινητοποιηθούμε και εμεί και οι λοιποί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο για την σωστή παρακολούθηση των κονδυλίων, γιατί θα έχουμε ζητήματα για διάφορε γραμμέ του προπολογισμού. Το νωρίτερο δυνατό λοιπόν να έχουμε αυτή την παρακολούθηση για να πιάσουν το από τα λεφτά μα. Η κυρία, πώ τη λένε αυτή την σοσιαλίστρια που πάντοτε μιλάει για τα λεφτά που πρέπει να πιάνουν τόπο. Αυτή, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα βρει την κατάλληλη απάντηση αν έχουμε την επιτήρηση εγκαίρω. Και επίση εθνικές δαπάνες και κράτη-μέλη, αναφέρθηκαν νωρίτερα. Ίσως θα πρέπει να αναστήσουμε, με δική μας πρωτοβουλία, τις ε, συνεδριάσεις. Ε, Παραδείγμα, την έχουμε μια συνάντηση μεταξύ Επιτροπής των Προπολογισμών και αντίστοιχων ε, εκπροσώπων των εθνικών, των κρατών μελών, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να λάβετε εσείς αυτή την πρωτοβουλία για να δούμε και οι δημοσιονομικοί μηχανισμοί τι θα επέτρεπαν για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων για να μην ε, θεωρήσουν αυτά ότι τα έχουμε αποκόψει από τη διαδικασία. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση προσθέτω στα όσα υπόθηκαν. Θα παρακαλέσω τον στο αλλά και τον Ράιμερ Μπέγκε να κοιτάξουν το κείμενο του ψηφίσματος του 2010. Ο Ράιμερ μπορεί στο έγγραφο εργασία του να αναφέρεται σε αυτό το σημειολογικό ζήτημα τι εστί ε, αναθεώρηση και τιμή και με κάποιες από τις ε, τροπολογίες μας προσπαθούμε να το διευκρινίσουμε το θέμα αυτό. Οι τροπολογίες 3, 4 και 5 συγκεκριμένα δικέ, μας πιστεύω καλύπτουν το θέμα γιατί ε, επανεξετάζουμε όλη τη διατύπωση και το τι θα πρέπει να γίνει για την περίοδο 2011-2013 και σημειώνουμε ότι αυτό στο οποίο προβαίνουμε δεν είναι απλώς μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση, αλλά τροποποιούμε και τα κονδύλια, τα ποσά δηλαδή όταν βλέπουμε ζητήματα στους διάφορους τίτλους. Και μετά, επόμενο στάδιο, τα όσα ακολουθούν από το 2013 και μετά. Παρακαλώ λοιπόν και τον Ράιμερ και τον Άσολο να το κοιτάξουν πολύ προσεκτικά αυτό το οποίο έχουμε προτείνει με τις τροπολογίες. Είναι πολύ σημαντικό με το ψήφισμα του 2010 να ξεκινήσουμε και να λέμε ξεκάθαρα αυτό το οποίο ε, θέλουμε. Με την ίδια διατύπωση που έχουμε ακολουθήσει για, το, για την πρόταση του 2010, για τον προπολισμό του 2010, όπως και για την έκθεση του κ. Έλλης. Ναι, τροπολογίες 3 και 4 λέει ο πρόεδρος. Και 5, και 5, ναι. Δύο λόγια, αν μου επιτρέπετε, πριν να ολοκληρώσω, Ρόιμερ, για να απαντήσω στον Τζέιμς. Είναι πολύ εύστοχη η ερώτησή σου, όντω. Τέτοιου ερωτήσει θα πρέπει να διατυπώσουμε προ τον υποψήφιο επίτροπο και σε όλου του υποψήφιου επιτρόπου. Το προτινόμενο κοινό ερωτηματολόγιο έχει ερωτήσεις του τύπου «Είστε έντιμος άνθρωπος» Ε, τι σας κάνει να πιστεύετε ότι είστε ικανός για τη θέση αυτή και άλλο τέτοια ερωτήματα. Αυτά που <laughs> πρέπει να απαντάει κανείς όταν συμπληρώνει την αίτηση βίζας για τις ΗΠΑ. Πολιτείες. Είσαστε κακό άνθρωπο, έχετε υπετιότητα για το ολοκαύτωμα, έχετε υπετιότητα για τον πόλεμο και διάφορα τέτοια πράγματα. Εξαίρετα, εξαίρετα, υπέροχα. Εν πάση περιπτώσει, τα ερωτήματα που συζητούμε εμεί τώρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύστοχα. για την ιδέα αυτή στην οποία αναφέρθηκε και στην οποία έχει αναφερθεί και η Κόζα επαναλημμένω. Θα ξέρει ασφαλώ ότι η Επιτροπή των Προπολογισμών κατόπιν πρότασή μου αποφάσισε να αναθέσει την ε, δεξαγωγή εκθέσεω για του προπολογισμού των κρατών μελών, έτσι ώστε να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση για ετήσιε συνεδριάσεις των Επιτροπών Δημοσιονομικών, των Επιτροπών ε, Προϋπολογισμών για να παρακολουθούμε την εξέλιξη των προϋπολογισμών μας και ταυτόχρονα μαζί με τον κοινοτικό προϋπολογισμό να κοιτάμε το κάθε κράτος μέλος μέσα στον προϋπολογισμό του να λαμβάνει υπόψη και τους κοινού ευρωπαϊκούς στόχους, να φροντίζουμε για να καλύπτεται και αυτή η διάσταση. Θα μπορούσαμε να το έχουμε και για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Δεν προβλέφθηκε, γι' αυτό είναι και ένας λόγος για τον οποίο να πέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της κρίσης του σχεδίου ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της κρίσης. 200 δισεκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκαν σε επίπεδο Συμβουλίου, 5 δις από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά εν τέλει δεν ξέρουμε τι έχει γίνει σε επίπεδο κρατών μελών για το σχέδιο ανάκαμψης και ο πρόεδρος Φαντρόμπο επιπλέον θα μπορούσε να αναλάβει την πρωτοβουλία μέσα από τα νέα του καθήκοντα και να προτείνει σε μια προσεχή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να λογοδοτήσει, να εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει, τι έχει δαπανίσει για να αντιμετωπίσει την κρίση. Αυτά τα 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποιο βαθμό τα απορρόφησε και με ποιο στόχο. Άρα πιστεύω θα πρέπει να είμαστε θέσει να διατυπώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Εμένα αυτές οι πρωτοβουλίες με βρίσκουν σύμφωνο. Θεωρώ ότι δεν απαιτούν νομική βάση, αρκεί πολιτική συμφωνία και νομίζω ότι με αυτή τη λύση μπορούμε να προχωρήσουμε αρκετά στον τομέα αυτό. Ράιμερ, θέλεις να απαντήσεις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή είχε προβλεφθεί η προσεχή συνεδρίαση τη Επιτροπή των Προπολογισμών ε, μόνο για τον Ιανουάριο, είχα ζητήσει να παρουσιάσω εγώ το έγγραφο από τώρα για να συστήσουμε τι βασικέ δομέ, για να ε, συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί, να είμαστε έτοιμοι, χωρί να είμαι σε θέση να επισέλθω ακόμη σε λεπτομέρειε, αλλά να έχω μια γενική επισκόπηση. Επισκόπηση και βέβαια έτσι να ξεκινήσουν και οι διμερεί επαφέ και με τι ομάδε και με του σκιώδει ηγητέ, του ταινιστέ των ομάδων. Ευχαριστώ ιδιαίτερω και για την αναφορά στο πενταετές πλαίσιο, στο πενταετές περιθώριο, που είναι σημαντικός στόχος για μας, ο πενταετής προγραμματισμός, είναι ένας στόχος για μας, αδιαπραγμάτευτος. Το θέμα είναι πώς θα τον καταφέρουμε, πώς θα τον εξασφαλίσουμε στην πράξη. και εγώ θα έλεγα προσαρμογή, επαλήθευση, αναθεώρηση και ε, παράταση του δημοσιονομικού προγραμματισμού θα μας πήγαινε για τις προσεχείς δημοσιονομικές προοπτικές του 2020 με εκλογές το 2014 και το 2019 υπενθυμίζω. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη ε, χρονική περίοδο στον προγραμματισμό μας. Από ό,τι φαίνεται δε ως προς τη γλώσσα, ως προς τη διατύπωση ε, η έννοια review δεν έχει μεταφραστεί πάντοτε όπως πρέπει. Στα ισπανικά η παραδείγματι δεν έχει την έννοια του review αλλά του revision που θα σήμαινε αναθεώρηση κειμένου και όχι αναθεώρηση θέσεων. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να μπω στα χωράφια του Λάσλο, ως ηγητής ε, για το ψήφισμα, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να διατυπώσω την εξή πρόταση οι τροπολογίες 2, 3, 4 και 5 των σοσιαλδημοκρατών ασχολούνται με το θέμα αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι τροπολογίες, υπάρχουν και άλλες, στις οποίες ε, και πάλι, σε περαιτέρω παραγράφους, εμφανίζεται το ίδιο ζήτημα, η ίδια τοποθέτηση. Θα έλεγα λοιπόν να συντονίσουμε τη διατύπωση αυτή, έτσι, ώστε αυτά τα τρία στάδια που προβλέπονται, στις τροπολογίες 2 έως 5, 3 έως 5, να ε, ακολουθηθούν κατά τρόπο πάγιο στο κείμενο. Ε, δεν έχω αντίρρηση αυτό δηλαδή, Απλώ θα ήθελα να μην έχουμε επικάλυψη και να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τα ίδια πράγματα. Θα πρέπει να γίνει προσαρμογή και ίσως θα μπορούσαμε, επί παραδείγματι, να πούμε στα αγγλικά, μαζί με την αναθεώρηση του σχεδίου για το 2011 έως 2030, επί παραδείγματι. Και εκεί Δεν ξέρω αν ο ή οι διαπραγματευτέ μπορούν να βρουν μια λύση, αλλά πάντω θα μπορούσαμε να βρούμε μια διατύπωση η οποία θα λέει ότι μιλούμε για την απαραίτητη προσαρμογή, adjustment, ανάλογα με τις εξελίξεις τη συνθήκη. Και εκεί μπορούμε μεταξύ μας οι ομάδες να βρούμε τη λύση και να μιλήσουμε για adjustment, review and revision, προσαρμογή, αναθεώρηση και επαναδιατύπωση, revision, του ε, πακέτου. Οπότε έχουμε καλύψει το σύνολο μέχρι, το, ε, μέχρι και το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα σε συμφωνία ελπίζω μεταξύ όλων των ομάδων. Έχουμε καλύψει τις έννοιες, τις έχουμε συμπληρώσει και έτσι ανταποκρινόμαστε και στα αιτήματα της τροπολογίας παριθμών 4 και μπορούμε να υποβάλουμε ένα πακέτο συνολικό στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων, στην Επιτροπή και το Συμβούλιο αν έχουν την καλοσύνη ο συγητή και οι σκιώδει να εξετάσουν αυτή την πρόταση και αν τους φαίνεται σκόπιμη να την ξαναδούμε και αύριο. Μπορούμε πάλι αύριο να το συζητήσουμε αν θέλετε. Κατά τα άλλα, θα πρότεινα πριν ακόμη από τις διακοπές των Χριστουγέννων να έλθει όποιο συνάδελφο ε, ενδιαφέρεται να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και διμερώ ακόμη. Εγώ πάντοτε προσπαθώ να διατηρώ και να, ε, να βρίσκω και το χρόνο και για τη συζήτηση βέβαια με του συντονιστέ. Αλλά είμαι διατεθειμένο οποιοδήποτε συνάδελφο έχει κάποια παρατήρηση να δεχτώ και να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ράιμερ. Καλώ. Λοιπόν, προτείνω να σταματήσουμε εδώ τη συνεδρία της Επιτροπής των Προπολογισμών και να επανέλθουμε αύριο το πρωί στις με τις ψηφοφορίες. Παρακαλώ να είμαστε όλοι παρόντες αύριο για την ψηφοφορία και να μείνουν οι συντονιστές. Ίσως και ο Ράιμερ αν θέλει ή αν χρειάζεται για να εξεταστεί για να εξεταστούν οι τροπολογίες του να ενδιαφέρουν περισσότερο. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, αντίρρηση. Ο Λάσλο, ο Βλαδίμιρ Μάνκα, οι συγητές επίσης, εάν το επιθυμούν, από τους λοιπούς συναδέλφους ε, δεν έχω παρά να ευχηθώ, να ευχαριστήσω καταρχάς ε, που θα αποχωρήσουν ταχύτατα από την αίθουσα και να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους. Σκεφτείτε ότι έπιασε πυρκαγιά ξαφνικά και χτυπάει ο συναγερμός. Φύγετε γρήγορα και ησύχως. Θα σας ξαναδούμε αύριο το πρωί.